Colleagues, please be seated. Ladies and gentlemen. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, κυρίες και κύριοι. Ώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μέρα της ε, συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ασφάλειας ε, και Άμυνας. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην ημερησία διάταξη και επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω σχετικά με την αποστολή της ΣΕΝΤΕ στην Ουκρανία. Στο Κίεβο και στην Ανατολική Ουκρανία συγκεκριμένα. Έχει γίνει παράδοση η υποεπιτροπή να πραγματοποιεί τέτοιες αποστολές. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Τέσσερις ευρωβουλευτές συμμετείχαν. που επισκέφτηκαν ε, και την πρωτεύουσα και την Ανατολική Ουκρανία. Εγώ ήμουν επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας αυτής. Επίσης συμμετείχε ο κύριος Γκάλερ από το ΕΛΚ, ο κύριος Γιάρομιρ Στετίνα, αντιπρόεδρος της ΣΕΝΤΕ και τελευταίος και καλύτερος ο κύριος Άρνε Λίτς από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Έχει γίνει η παράδοση να ξεκινάμε τις αποστολές με ενημέρωση και ανταλλαγή ε, απόψεων ε, με τους επικεφαλείς ε, της κοινότητας των Τατάρων της Κρυμαίας τον κύριο Μουστόφα Τζεμίλεφ συναντήσαμε, που είναι ο μυθικός ε, πια ηγέτης των Τατάρων της Κρυμαίας. Ε, συναντήσαμε και τον κύριο Τσπάροφ. είναι ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου των Τατάρων της Κρυμαίας ε, που έχει κηρύξει παράνομο ο, ε, ο Πούτιν. Συζητήσαμε την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, συζητήσαμε τους εξοπλισμούς. Συζητήσαμε την ε, πολύ ανησυχητική προοπτική του να υπάρχουν στην Κρυμαία στρατηγικά όπλα. Ενημερωθήκαμε επίσης ε, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εκφοβισμό της κοινότητας των Τατάρων και Ουκρανών και συζητήσαμε και την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια. Μετά από επίσκεψη στην θάλασσα Αζόφ, και την ε, ολοκλήρωση της γέφυρας στο Κέρτς. Δύο σημαντικές συναντήσεις είχαμε στα κεντρικά γραφεία του UAM με τον κύριο Ρόμαν Τρούμπα που είναι επικεφαλής του Γραφείου Ερευνών και μας ανέφερε διάφορα προβλήματα. Ελπίζω οι συνάδελφοι να αναφερθούν ε, εκτενέστερα σε αυτά. Ως συνήθως, είχαμε και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λατσίνσκας. και είχαμε μια σειρά συναντήσεων μαζί του. Επίσης, μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με την οργάνωσή του και εδώ στις Βρυξέλλες. Είχαμε μια ολόκληρη μέρα στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της οποίας λάβαμε εκτενή ενημέρωση από τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο. Συναντήσαμε τον αναπληρωτή υπουργό άμυνας ε, για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ε, και τον ε, Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας. Συναντηθήκαμε επίσης με σημαντικά μέλη του Κοινοβουλίου, Ράντα, Συναντήσαμε την κυρία Χάνα γραμματέα της Επιτροπής Ασφαλείας του Κοινοβουλίου. Επίσης, την δεύτερη μέρα μετά την επιστροφή μας από την Ανατολική Ουκρανία, τη μέρα αυτή την περάσαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Γνωρίζετε ότι είναι σημαντική προσωπικότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, παρακολουθήσαμε ε, μια σημαντική ομιλία του Προέδρου στο Κοινοβούλιο, Φερχόφνα Ράντα, σχετικά με αλλαγές στο Σύνταγμα. καθώς ε, και γνωρίσαμε επίσης ε, και συναντήσαμε μάλλον και την Υπουργό, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά, διότι ε, έχει μιλήσει και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ εδώ στο Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την Ανατολική Ουκρανία, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τις Ουκρανικές αρχές που μας βοήθησαν όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς. Χωρίς την ε, βοήθεια αυτή δεν θα, θα τα είχαμε καταφέρει, διότι έπρεπε να καλύψουμε μεγάλη απόσταση. Με ελικόπτερα, λοιπόν, μας μετέφεραν. Ξεκινήσαμε τις συναντήσεις μας στην Μαριούπολη, όπου ενημερωθήκαμε από το Ανατολικό Κυβερνείο των ε, ενόπλων δυνάμεων στην Μαριούπολη. Ήταν ε, εκτενής ενημέρωση, ενημερωθήκαμε για θέματα ασφάλειας. Καλωσορίζω και τον προσκεκλημένο μας, ε, τον κύριο Γελισέη, που ήταν ε, πρέσβης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον βλέπαμε τακτικά στο παρελθόν. Τώρα πια είναι αναπληρωτής προϊστάμενος του Περιοδικού Γραφείου. Επισκεφτήκαμε το Τόρσκ. μάλλον όχι, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Μαριούπολη. Ενημερωθήκαμε όχι μόνο για την ασφάλεια και την άμυνα, συναντήσαμε και την ε, τοπική κυβέρνηση, το Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης, ε, τους αναπληρωτές δημάρχους, και συζητήσαμε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της περιοχής. Συζητήσαμε προκλήσεις και κινδύνους που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό ε, λιμένων. Κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ήταν ε, μακρά η συζήτηση, όλο το βράδυ κράτησε και νομίζω ότι ενημερωθήκαμε καλά σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας εκεί, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών ως προς τις μεταφορές, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Μαριούπολης και τον αποκλεισμό λιμένων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί δυσκολίες και όσον αφορά τη διαχείριση της περιοχής και όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξή τη. Επισκεφτήκαμε στην Ταλακίφκα το σχολείο, βρίσκεται κοντά στη Μαριούπολη και χρηματοδοτείται το σχολείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επόμενη μέρα ταξιδέψαμε με ελικόπτερο στο Κράματόρσκ. και επισκεφτήκαμε τους ειδικού παρατηρητές του ΟΑΣΕ και θα έπρεπε να αναφέρω ότι και στο Κίεβο συναντηθήκαμε με τον πρέσβη Σάιντικ που μας ενημέρωσε σχετικά με την όλη αποστολή του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία, καθώς και πολιτικά, διαδικαστικά και πρακτικά θέματα. Uh, Στο Κραματόρσκ Είχαμε μία μάλλον σύντομη συνάντηση. Έπρεπε να βιαστούμε να συναντήσουμε εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και από τις δύο πλευρές. Και ε, μετά φτάσαμε στο πέρασμα προς το Μαγιόρσκ. Δεύτερη φορά επισκέφτομαι εγώ προσωπικά το μέρος αυτό. Ήμουν εκεί και πριν από ένα χρόνο. Έτσι μπόρεσα με τα ίδια μου τα μάτια να διαπιστώσω τις εξελίξεις. Είδαμε ότι και η, αυτή η ύφκα έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί, αλλά υπό ε, πολύ κακές συνθήκες. Και τα κτίρια βρίσκονται σε κακή κατάσταση και οι προμήθειες ε, είναι ισχνές. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση της ε, αξιολόγησης της κατάστασης της ασφαλείας στην περιοχή αυτή. Αυτά σε συνάντηση με ε, στρατιώτες και αξιωματικούς στην Αντιγεύκα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επισκεφτούμε το Z-Point, ο κ. Στρεβίτσιους, πρόεδρος ε, των φίλων της Ουκρανίας, επισκέφθηκε το σημείο αυτό πέρσι, αλλά μάθαμε ότι υπήρξε ένα περιστατικό στην Μαγιόρσκ μετά από την παραμονή μας εκεί και γι' αυτό δεν καταφέραμε να επισκεφτούμε αυτό το σημείο της γραμμής που περνάει από την Αυτιγίφκα. Από την Αυτιγίφκα πήραμε το τρένο για το Κίεβο ε, και σας ενημέρωσα ήδη για τις συναντήσεις που είχαμε στο Κίεβο. Αυτή λοιπόν ήταν η δική μου ενημέρωση. Ο κύριος Γκάλερ, παρακαλώ όχι, ο κύριο παρακαλώ. Δεν θα ήθελα να τονίσω πολλά περισσότερα. Να πω ότι πρέπει να δείξουμε την παρουσία μας ειδικότερα στην Ανατολή για να δούμε τον αντίκτυπο της επιθετικής συμπεριφοράς της Ρωσίας εκεί. Και στο Κίεβο θα δείξουμε έτσι, αλλά και σε όσους είναι ενεργοί εκεί από κοινού τον ε, ΟΑΣΕ και άλλους ε, να, δούμε, να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, προσπάθειά της να βοηθήσει την Ουκρανία, ειδικότερα στην ανατολική πλευρά της, εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Νομίζω ότι το να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα είναι σημαντικό. Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης και άλλοι θύνοντες εκεί Μα ζήτησαν ε, στο Κίεβο επειδή ο κύριος Γέλτσιεφ είναι εδώ, ε, θα ήθελα να το επαναλάβω, μας είπαν παρακαλώ ξανανοίξτε το αεροδρόμιο στη Μαριούπολη. Ξέρουμε βέβαια ότι είναι πολύ κοντά στο ε, σύνορο και αυτό είναι το επιχείρημα. Ε, παρόλα αυτά όμως δεν θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική αεροπορία εκεί ε, ή θα ήταν μια τεράστια οικονομική όθηση για την περιοχή το να ξανανοίξει το αεροδρόμιο της Μαριούπολης και νομίζω ότι ε, παρά την πτώση του αεροσκάφους που είχε γίνει εκεί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα αέρια ασφάλεια επαρκή στην περιοχή. Αυτό ακριβώς ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουν την υποστήριξη από μας ε, ε, στην κοινωνία των πολιτών όλοι όσοι εμπλέκονται στην περιοχή και προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να επενεθεί το έργο τους για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερότερη κατάσταση στην περιοχή. Ο κύριος Στέτινα Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, επειδή θα μιλήσω τσεχικά, βάλτε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα πολύ σύντομα να επωφεληθώ της ευκαιρίας ε, για να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο ε, για την ενημέρωση θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω του, τη Γραμματεία και όλους όσους υποστήριξαν γραμματιακά αυτήν την αποστολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τον Ουκρανικό στρατό που μας βοήθησε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που είχαμε εγκρίνει. Το πιο σημαντικό τμήμα του προγράμματος ήταν η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του Ουκρανικού στρατού που μας ενημέρωσαν για την κατάσταση στη θάλασσα του Αζόφ που είναι κάτι που θα συζητήσουμε με τον κύριο πρέσβη Γελίσιεφ. Πρέπει λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το ε, θέμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που η κυρία Φωτίγκα, η πρόεδρος της Επιτροπής μας, ε, το είχε θέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, κατά ε, κατά την ενημέρωσή μου. Ξέρετε ότι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας έχει άμεση σχέση με αυτό το, με τη σημασία της παρουσίας μας για λόγους ασφαλείας στην περιοχή, η κατάσταση της ασφάλειας ε, στη θάλασσα του Αζόφ ήταν ένα θέμα που μας απασχολούσε πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Στετίνα ότι η ενημέρωση που λάβαμε από το αρχηγείο της ε, Ουκρανίας ε, για την ανατολική περιοχή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και πραγματικά όλος ιδιαίτερος την εκτιμούμε. Να περάσουμε τώρα, δεν υπάρχουν περισσότερες παρατηρήσεις, πλέον παρατηρήσεις για την ενημέρωση αυτή, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η εξελίξη στην κατάσταση ασφάλειας της θάλασσας του Αζόφ. Με χαρά Θα ε, καλωσορίσω τους τρεις ε, εξέχοντες ομιλητές μας, ε, τον Λουκ Ντεβίνια, τον γνωρίζετε πολύ καλά, είναι αναπληρωτής διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα γνωρίζετε βεβαίως τον πρέσβη Κωνστιαντίν Γελισέγεφ, Παραμένετε πρέσβης. Είστε αναπληρωτής προϊστάμενος του Προεδρικού Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Καλώς ήρθατε. Και είναι εδώ μαζί μας και η κυρία Ραντοσουάβα Στεφάνοβα που είναι η προϊσταμένη του τομέα Ρωσίας και Ουκρανίας στη μονάδα πολιτικών υποθέσεων και πολιτικής ασφάλειας στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Όχι μόνο λόγω της αποστολής ε, στην ε, Ουκρανία, αλλά επειδή παρακολουθούσα την κατάσταση της ασφάλειας ε, στη θάλασσα του Αζόφ ε, εκ του από προσωπικής μου εμπειρίας και για λόγους προσωπικού ενδιαφέροντος για πολλά χρόνια στη λίμνη Βιστούλα μακριά Ε, επειδή εγώ μεγάλωσα στην Πολωνία σε ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μπλόκαραν οι Ρώσοι ε, με παρόμοιες ε, ενέργειες με αυτές τις οποίες προβαίνουν σήμερα. Άλλαξε όμως η κατάσταση όταν εμείς στην Πολωνία και μάλιστα εγώ είχα το προνόμιο να ήμουν μέλος της κυβέρνησης εκείνη την εποχή αποφασίσαμε να υπάρξει ένα ένα διάβλο για να μπορέσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μπλοκάρισμα της Ρωσίας Φυσικά είναι διαφορετική η δυσκολία της κατάστασης. Δεν λέω ότι μπορούν να συγκριθούν. Ε, πάντως, όταν μίλησα με μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Μαριούπολης και μου είπαν ότι όταν πολλά χρήματα ε, διατίθενται, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και αυτό συμπεριλαμβάνει βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας από τους ε, μεγαλύτερους δωρητές στην περιοχή. Ε, σε πολύ δύσκολα σημεία μπορούμε να μπλοκάρουμε την δυνατότητα μεμονωμένων εξελίξεων στην περιοχή και πράγματι το είδαμε αυτό επιχειρηματικές δεξιότητες ε, απλών ανθρώπων στο ανατολικό τμήμα της Μαριούπολης και πιστεύω ότι με τις απαραίτητες ε, ε, συνθήκες η Ουκρανία μπορεί πραγματικά να αναπτυχθεί, οι Ουκρανοί μπορούν να αναπτυχθούν από μόνοι τους και να είναι ένας ισότιμος εταίρος για όλους μας. Η κατάσταση της ασφάλειας όμως πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου, όχι μόνο λόγω της ε, προσάρτησης της Κρυμαίας, με τις πολύ κακές συνέπειες που είχε αυτό, ε, για στρατηγικούς, ε, στρατιωτικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας, για όλους μας, όχι μόνο για την Ουκρανία. όχι μόνο στην ε, Βαλτική, αλλά και πέρα από αυτήν, υπάρχουν τώρα περαιτέρω εξελίξεις, γιατί χτίζεται μία γέφυρα πάνω από το στενό του Κέρτς, και αυτό το μπλοκάρισμα, ε, της, η απομόνωση των ε, λιμανιών στη θάλασσα του Αζόφ θα επηρεαστεί βεβαίως. Έχετε το λόγο κύριε Ντεβίνια. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ε, καλημέρα σας. Θα ήθελα να, καλώς, να χαιρετήσω και τους συναδέλφους. Είναι μεγάλη χαρά να μιλώ σήμερα για ένα θέμα το οποίο είναι στο επίκεντρο και ε, μεταξύ των προτεραιοτήτων της εξωτερικής μας πολιτικής να πω καταρχάς ότι παρά το γεγονός ότι ακούμε συχνά φωνές που λένε ότι η κρίση ε, στην Ουκρανία έχει ξεχαστεί ή ότι η διεθνής προσοχή θα έπρεπε να εστιαστεί σε άλλα ε, θέματα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Για μας η εξωτερική πολιτική παραμένει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό για την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας ε, και αυξάνεται συνεχώς ε, η ενίσχυσή μας επειδή η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις. Είναι λοιπόν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας, ε, του θεματολογίου μας, στο, στις συζητήσεις του Συμβουλίου με τα κράτη-μέλη, όπως επίσης και σε σχέση με την ανανέωση των σχετικών κυρώσεων. Ε, ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει και στα διεθνή φόρα που συζητούν το θέμα. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, ε κάποια κόποση που να έχει επέλθει από τη συζήτηση αυτού του θέματος. Μετά την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας λόγω της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία, η κατάσταση στην θάλασσα του Αζόφ ε, επιδεινώθηκε. Είναι μια πολύ, ένα πολύ περίπλοκο πλέον ε, περιβάλλον ασφαλείας και φυσικά επειδή θα γίνει πάνω από την χερσόνησο της Κρινέα στο στενό του Κέρτς μια καινούρια γέφυρα υπάρχουν νέα ζητήματα όσον αφορά την κυριαρχία της Ρωσίας συγγνώμη, της Ουκρανίας, λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Ε, υπάρχει μία απομόνωση της περιοχής από την Ουκρανία, ε, στην οποία ανήκει, υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί που τίθενται στα σκάφη που περνούν από αυτό το ε, στενό, κάτι το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ουκρανική οικονομία. Από το Μάιο δυστυχώς έχουμε δει ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να, ε, να εφαρμόζει ένα νέο καθεστώς επιθεωρήσεων ε, στο Περδιάνσκ και στη Μαριούπολη. Αυτές οι επιθεωρήσεις που είναι καταχρηστικής φύσεως παρεμποδίζουν ε, το, το πέρασμα των πλοίων και δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις, κάτι το οποίο έχει αυξήσει το κόστος των μεταφορών. Και έχουμε δει ότι οι επιθεωρήσεις έχουν ε, αυξηθεί από δύο ώρες πριν από μερικούς μήνες σε τρεις μέρες προσφάτως. Οπότε ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο τα ουκρανικά σκάφη και την ουκρανική οικονομία αλλά και για τα ε, σκάφη της Ένωσης και τις οικονομίες τους ε, γιατί υπάρχουν 20-30 σκάφη που περιμένουν ανα πάσα στιγμή να γίνουν αυτές οι καταχρηστικές επιθεωρήσεις. Η Ρωσία έχει συνεχίσει την στρατιωτικοποίηση της θάλασσας του Αζόφ και μας απασχολεί πάρα πολύ η ανάπτυξη των ε, ε, δυνάμεων στην περιοχή, σε μια περιοχή η οποία ήταν ε, σχεδόν πλήρως αποστρατικοποιημένη. Οι αναλυτές λένε ότι ο στόχος είναι της Ρωσίας να, να ελέγχει την πρόσβαση στη θάλασσα του Ασόφτου. Το 2003 υπήρχε μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρουσίας για αυτό το συγκεκριμένο σημείο και ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διαβουλεύσεις σε περίπτωση προβλημάτων και διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να χαιρετήσω την πολιτική της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει κατά το μέγιστο διπλωματικά μέσα όσο χρειάζεται αυτό ε, και βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν ε, νομικά μέσα ε, στο Διεθνές Δικαστήριο όπως για παράδειγμα υπό τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ στο Διετητικό Δικαστήριο. Όσον αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουμε ότι αντιδράσαμε πολύ γρήγορα, Εξετάσαμε την ε, ε, κατασκευή αυτή τη γέφυρα χωρί τη συγκατάθεση τη Ουκρανία και εκφράσαμε τι βαθιέ μα ανησυχίε για την επιδείνωση τη κατάσταση και στον Εύξηνο ε, Πόντο και σε άλλε θάλασσε. Ε, όπως γνωρίζετε, στις 31 Ιουλίου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε τρεις ε, ε, εταιρείε που συμμετείχαν στην κατασκευή της γέφυρας σε περιοριστικά μέτρα, γιατί θεωρεί ότι απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. θα ήθελα να πω η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεπισημαίνει την υποστήριξή της στην Ουκρανία, το έχουμε εκφράσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και τη δεσμευσή μας να την υποστηρίξουμε, όπως έγινε και στην πρόσφατη σύνοδο ε, την περασμένη εβδομάδα, στην ε, ε, σύνοδο σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ε, κύριε Γελισιέιεφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φωτίγκα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και χαίρομαι και για την παρουσία του φίλου μου του Λουκ Ντεβίν και ευχαριστώ και την κυρία Στεφάνοβα. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε άλλο ένα σημείο ένταση στην επικράτεια της Ουκρανίας μετά από που δέχεται ρωσική επίθεση αναφέρθηκε από τις 29 του Απρίλη φέτος με την δημιουργία της γέφυρας η Ρωσία άρχισε να μπλοκάρει ενεργά τη διάλευση των εμπορικών σκαφών στην θάλασσα του Αζόφ που πηγαίνουν στον Περκάνσκι και στη Μαριούπολη. Η παραβίαση λοιπόν του τη ελεύθερη διέλευση που διασφαλίζεται από το Διεθνές Δίκαιο τη θάλασσα και το Διεθνές Δίκαιο και από διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας Ουκρανία, ήδη αφορούσε γύρω στα 300 πλοία και τα περισσότερα από αυτά είχαν σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ήδη ανέφερε ο Λουκ. Μιλάμε για χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, Καναδάς, ε, Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος, ε, κατοχώρες, Ρουμανία, Τουρκία. Πολλά από αυτά λοιπόν έγιναν πολύ κοντά στις Ουκρανικές ακτές παρά τα ισχύοντα σε σχέση με τα μίλια από την ακτή. Είχαμε πολύ ενδελεχείς ελέγχους, όπως θα τους έλεγα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Ξέρετε ότι η Ρωσία ξεκίνησε το χτίσιμα του φράγματος στο νησί Τούσλα το 2003, ακριβώς για να τιμωρήσει την Ουκρανία για τα πρώτα βήματα τότε που έκανε προς την ανεξαρτησία της, προς την Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και το 2014, με την επέμβαση την αιματηρή στην Ουκρανία, τιμωρούσε την Ουκρανία για την συμφωνία σύνδεση και τώρα επιτίθενται στην θάλασσα του Αζόφ. Και η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη αν δούμε ακριβώ και τι στρατιωτικέ πτυχέ. Εκτό από μια μεγάλη κλίμακα στρατιωτικοποίηση τη Κρυμαία, η οποία ήδη αναφέρθηκε, μπαίνει πια μυστικό, η Ρωσία άρχισε να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην θάλασσα του Αζόφ, η οποία ήταν αποστρατιωτικοποιημένη. Η Ρωσία κοντεύει, ολοκληρώνει τις δράσεις της στη θάλασσα του Αζόφ. Θέλουν να φτιάξουν μια νέα στρατιωτική βάση με τη μεταφορά θεωτικού υλικού από την Κασπία. Μαζί με τις δραστηριότητες βέβαια της ακτοφυλακής και του ρωσικού ναυτικού στην Μαύρη Θάλασσα, όλα αυτά και στη θάλασσα του Αζόφ. Επίσης, η ε, κοντά στη Φεντόσα ε, έχουμε μεταφορά όπλων με πυρηνικές κεφαλές από τη Ρωσία. Με αυτή την τακτική η Ρωσία θέλει να πετύχει τους εξής στόχους. Πρώτον, χρειάζεται ένα διάδρομο για την ε, κατεχόμενη Κρυμαία. Θέλουν να περικυκλώσουν τις Ουκρανικές δυνάμεις μέσω της παρουσίας τους στη θάλασσα του Αζόφ για να αποφύγουν ακριβώς χερσέ ε, ε κινήσεις οι οποίες είναι πολύ ακριβές για αυτούς. Η Μαριούπολη και άλλες τοποθεσίες είναι ακριβώς τεράστια σημασία για την Ουκρανική βιομηχανία και η Ρωσία πιστεύει ότι οι χιλιάδες ανέργων αποτελεί ένα, μια ευκαιρία για αυτούς. Και όπω είπε και η κυρία Φωτήγα προηγουμένω, ίσω θα έπρεπε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πώ θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτή ακριβώ την περιοχή, για τον Μπεργκάντ και τη Μαριούπολη, κοινωνικών και οικονομικών προγραμμάτων αποκατάσταση αυτών των περιοχών, ώστε ακριβώ να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ανέργων, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική κατάσταση σε αυτήν την τόσο σημαντική στρατηγική περιοχή, θα έλεγα. Στόχοι λοιπόν της Ρωσίας. Η Ρωσία χρειάζεται ένα απόλυτο έλεγχο στην θάλασσα του Αζόφ και στη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτός ο έλεγχος θα δώσει την ευκαιρία στη Ρωσία να αποσταθερήσει περισσότερο την Ουκρανία, την Νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, να παρακάμψει το, την αστερό πλευρό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην θάλασσα του Αζόφ νομίζω η Ρωσία δοκιμάζει τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημοκρατικής κοινότητας. Βεβαίως, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, χώρες μέλη που είναι στο ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την επιθετική αυτή συμπεριφορά λόγω ακριβώ τη τάση του στη θάλασσα του Αζόφ. Επίση, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλου εταιρού, χώρε εταιρού, να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα κατά των λιμένων της Ρωσίας στη θάλασσα του Αζόφ. Επειδή η Ρωσία χρησιμοποιεί τα λιμάνια αυτά για να παραβιάσει ακριβώς τις κυρώσεις της Ένωσης. Γι' αυτό κατά την άποψή μας ελπίζουμε ότι αυτές οι κυρώσεις θα θεσπιστούν κατά των ρωσικών στη θάλασσα του Ασόφ. Επίση, δοκιμάζουν αυτέ τι στρατιωτικέ τακτικέ που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν σε άλλε περιοχέ, στην Βαλτική, στη Μεσόγειο. Αποτελεί δηλαδή ένα είδο προημίου για επερχόμενες μελλοντικέ στρατιωτικέ κινήσεις. Έχουμε ασκήσει ασκήσεις κοντά στην οικονομική ζώνη τη Σουηδίας και τον Απρίλιο είχαμε ε, δοκιμές πυράβλων από τη Ρωσία ε, πολύ κοντά στην Λετωνία χωρίς, χωρίς να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας. Με αυτές λοιπόν τις παράνομες δράσεις η, στη θάλασσα του Αζόφ και αλλού η Ρωσία δεν τηρεί, ακριβώς δεν τηρεί κανένα α, διεθνή κανόνα και αυξάνει την επιθετικότητα και την όρεξή της για περαιτέρω παράνομες δράσεις. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιθετική στάση και ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχάς με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα. Ξέρετε ότι ήδη στη θάλασσα του, θάλασσα του Αζόφη ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίε επιδιαιτησία ε, βασιζόμενοι στο δίκαιο της θάλασσας του 1982. Άγκλος. Επίσης, ελπίζουμε να προστατεύσουμε τα χωρικά μας ύδατα, την ανεξαρτησία μας και τα νομικά μας συμφέροντα συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συμφερόντων στην θάλασσα του Αζόφ. Παρ' όλα αυτά, εδώ δεν είμαι μόνο για να παραπονηθώ, αλλά για να στείλω και ένα μήνυμα στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ενεργοί, πιο αποφασιστικοί. Εμείς Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ισχυρές δηλώσεις υπέρ της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της, της Ουκρανίας, ιδιαίτερα για την Κρυμαία και θάλασσα του Αζόφ. Όμως θα πρέπει να τα φέρουμε αυτές τις καλές ισχυρές δηλώσεις στην πράξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράσεις και από τον ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως Είμαστε ευνόμονες και το ότι τις επόμενες εβδομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε μια ιδιαίτερη ακρόαση που θα αφορά τη θάλασσα του Αζόφ και καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από αυτές τις συζητήσεις να υιοθετήσει ένα πολύ ισχυρό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο ακριβώς θα καταδικάζει τις ρωσικές επιθετικές δράσεις και θα ζητά από το Συμβούλιο της Ένωσης να θεσπίσει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τώρα μιλάμε και βλέπετε εδώ για τη γέφυρα που λέγαμε ότι χτίζουν. Ήταν χαμηλού προφίλ η αντίδραση της Ένωσης για τη γέφυρα. Είχαμε κυρώσεις μόνο κατά έξι ρωσικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην στο χτίσιμο της γέφυρας. Αυτό όμως φίλοι μας δεν είναι τίποτα. Χρειαζόμαστε κάτι το πιο ισχυρό και όχι μόνο κάτι που να αφορά τις κατασκευαστικές. Να, να βάλουμε κυρώσεις και σε αυτές τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη γέφυρα. Μπορούμε να σας δώσουμε, αν θέλετε, έγγραφα, τεκμηρίωση κτλ. Μετά, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναθεωρήσει τις κυρώσεις κατά ε, και των ρωσικών λιμένων στη θάλασσα του Αζόφ. Και κάτι άλλο. Βασιζόμαστε, στηριζόμαστε στο γεγονό ότι κάποιες χώρες της Ένωσης θα σταματήσουν την στρατιωτική τεχνολογική συνεργασία με τη Ρωσία ώστε να υποβαθμίσουν την στρατιωτική συνεργασία με τα ρωσικά πλοία, γιατί δεν είναι μυστικό ότι κάποιε χώρε συνεργάζονται σε αυτό το τομέα με τη Ρωσία. Οπότε αυτό το είδο ε, συνεργασία θα πρέπει να σταματήσει αμέσω. Και βεβαίω στηριζόμαστε στην περαιτέρω συνεργασία με του εταίρου μα από το ΝΑΤΟ, την Ένωση και τη ΣΥΠΑ, ώστε να ενισχύσουμε τι ικανότητε τη Ρωσία μέσω του εξοχρονισμού του Ουκρανικού στόλου. Επίσης, θα θέλαμε να ενισχυθεί η δέσμευση συμμετοχή της Ένωσης στη Μαριούπολη και στο Τριάνσκ που όπως ανέφερα προηγουμένως θα μπορούσε να, θα να συμβάλλει η Ένωση με επενδύσεις, ε, με δράσεις για τη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης εκεί. Και βεβαίως, για να είμαι σύντομος, να σας πω ότι εμείς θέλουμε μία ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης, όχι μόνο στη θάλασσα του Αζόφ και στα στενά, αλλά και στον Ντόμπασκ. Ξέρετε ότι δυστυχώς η Ρωσία δυστυχώς συνεχίζει την επιθετική της πολιτική στην Ανατολική Ουκρανία και είχαν παραδείγματα των προθέσεων της Ρωσίας για διεξαγωγή νοθευμένων εκλογών τον Νοέμβρη στο Λογκάτσκ και στο Ντόνετσκ. Γι' αυτό ακριβώ καλούμε του εταίρου μας τη Ένωση όχι μόνο να καταδικάσουν αυτά, αυτά τα σχέδιά τους, αλλά να πούν ξεκάθαρα ότι αν αυτές οι εκλογές λάβουν χώρα, τότε η Ρωσία θα πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα. Τώρα, τι τίμημα είναι αυτό, τι να σα πω. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την επιθετικότητα της Ρωσίας μόνο μέσω παγκοσμίων κυπέλων ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Νομίζω μόνο με συγκεκριμένε πολιτικέ εκ μέρου τη Ένωση θα μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτή την επιθετική δραστηριότητα τη Ρωσική Ομοσπονδία. Γι' αυτό ακριβώ στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη τη Ένωση, στι σοφέ αποφάσει τη Ένωση σχέση με την φάση τη ε, επέκτηση και παράταση των κυρώσεων, αλλά νομίζω τέρμα τα λόγια θα πρέπει τώρα να αυξήσουμε το επίπεδο των κυρώσεων, λαμβάνοντα υπόψη όχι μόνο την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και την κατάσταση στην Σκατοχώρε, στο Σόλσπερι και σε πολλά άλλα μέρη. Φίλοι, σε σχέση με το Brexit, με την υπόθεση του Σόλσπερι, Κρυπάλ, με την περίπτωση με τα, χημικά της Ολλανδίας, όλα αυτά ξεκίνησαν από την Ουκρανία η δηλητηρίαση των, των ξεκίνησε από την Ουκρανία, όπου έφυγαν από εκεί και πήγαν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο περίπτωση των Ολλανδικών χημικών ξεκίνησαν από την ε, Ουκρανία, Κρυμαία κλπ. Συρία κλπ. Οπότε φτάνει πια. Υπάρχουν τεκμήρια, υπάρχουν αποδείξεις, οπότε η κυρώσει τη Ένωση και τη διεθνή κοινότητα θα πρέπει να ενισχυθούν. Και καταλήγοντα για άλλη μια φορά, να επαναλάβω ότι η έλλειψη αντίδραση οδηγεί στην κλιμάκωση τη κατάσταση εκ μέρου των δρόσεων. Θέλουμε ενότητα, αλληλεγγύη και μια κοινή απάντηση την καλύτερο τρόπο δηλαδή ώστε να κάνουμε τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνέ δίκαιο και την ε, εδαφική ακυρότητα τη χώρα. ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε η Ελισέγεφ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ραντοσλάβα Στεφάνοβα από τον ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω να μιλήσω εδώ. Βρίσκω πάντα θετικές τέτοιες συζητήσεις ανάμεσα στους οργανισμούς μας, αλλά και με τους ε, Ουκρανούς εταίρους μας. Πολλά υπόθηκαν ήδη από τους προλαλήσαντες. Εγώ θα επικεντρωθώ στην προοπτική του ΝΑΤΟ. Θα σας περιγράψω πώς βλέπουμε εμείς ε, την ε, κατάσταση ασφαλείας ε, στη θάλασσα του Αζόφ. Καταρχάς, από πλευράς των μελών του ΝΑΤΟ, θεωρούμε ότι η θάλασσα του Αζόφ συνδέεται στενά με την ασφάλεια στον Εύξενο Πόντο και στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κάτι που αφορά τη δική μας ασφάλεια. Γνωρίζοντας τις δράσεις που έχει αναλάβει το... Ε, που έχουν αναλάβει οι, δράσ... Ρώσοι, ε, αυτά αποτελούν το βασικό λόγο για τις δικές μας ενέργειες. Και έχουμε τρία μικρά κράτη του ΝΑΤΟ εκεί και έχουμε και άλλες χώρες εταίρους των οποίων η ασφάλεια συνδέεται με τη δική μας. Γι' αυτό, ήδη πριν δύο χρόνια, με την διάσκεψη της Βαρσοβίας ε, έχουμε εγκαθιδρύσει την δύναμη Τέιλοφόρντ στην πλευρά του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Και έτσι έχουμε πολυμερές στρατηγείο στην Ρουμανία. Επίσης έχουμε ενισχύσει την ενέργεια στην όμευση της περιοχής. Έχουμε αυξήσει και την παρουσία μας στη θάλασσα και έχουμε και περισσότερη συνεργασία με τους εταίρους μας, ιδιαίτερα με την Ουκρανία. Φυσικά, να πάσα στιγμή, οι ηγέτες μας ήταν διατεθειμένοι να εκφράσουν να καταδικάσουν τις δράσεις της Ρωσίας ε, και στον Ευσυνοπόντο και αλλού. Έχουν καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες αυτές ε, και εδώ στις ε, Βρυξέλλες τον Ιούλιο είχαμε μια δήλωση όπου καταδικάζεται η κατασκευή της γέφυρας. Παρακολουθούμε στενά οποιαδήποτε κλιμάκωση μπορεί να δημιουργηθεί από την ολοκλήρωση ή την ε, περαιτέρω οικοδόμηση της γέφυρας αυτής. Επίσης, έχουμε καταδικάσει την ε, στρατιωτικοποίηση ε, της περιοχής και ιδιαίτερα της θάλασσας του Αζόφ. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αποφάσεις και δηλώσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς. Πέρα από αυτό έχουμε ενισχύσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ιδιαίτερος εταίρος μας και ο πρέσβης Γελίσιεφ αναφέρθηκε στην βοήθεια που έχουμε παράσχει στη χώρα. Ιδιαίτερα έχουμε ενισχύσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να ανοικοδομήσει την ε, σημαντική ε, θαλάσσια δύναμή της που καταστράφηκε κατά την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας από την Ρωσία. Έχουμε λοιπόν εκφράσει την υποστήριξή μας προς την ε, Ουκρανία. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την προσάρτηση της Κρυμαίας από την ε, Ρωσία και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στην ε, αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής Ντονβάς. Θα ήθελα να σας περιγράψω τι κάνει το ΝΑΤΟ ιδιαίτερα στον θαλάσσιο τομέα για να στηρίξει την Ουκρανία. Ίσως όχι σε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε σημαντική παρουσία στο Κίεβο. Έχουμε τετραπλασιάσει το προσωπικό στο γραφείο μας εκεί, με εμπειρογνώμονες που δίνουν συμβουλές ε, για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα ασφαλείας. Έχουμε και συμβούλους σε διάφορους φορείς της Ουκρανίας, όπως είναι το Υπουργείο Αμήνης, και έχουμε συνεργαστεί στενά με στόχο την ε, ανάπτυξη του στόλου. Και αυτό είναι πολύ θεμελιώδες. Θέλουμε να βοηθήσουμε το ΝΑΤΟ ε, στην προσπάθειά του να προσφορήσει στην συμμαχία και έτσι θέλουμε ε, να τους μεταφέρουμε βέλτιστες πρακτικές ε, από την Ευρώπη και τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Για να βοηθήσουμε λοιπόν καλύτερα την Ουκρανία, πέρα από την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης ε, και νομικών συμβουλών, συνεργαζόμαστε στενά με το Κοινοβούλιο κατά την εκπόνηση νομοθεσίας. Είχαμε πρόσφατα τον νόμο για την εθνική ασφάλεια, τον οποίο επικροτούμε. Επίσης, συμμετέχουμε σε όλο και περισσότερες ασκήσεις με την Ουκρανία για να προωθήσουμε την διαλειτουργικότητα των δυνάμεών μας. Η Ουκρανία έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και στη θάλασσα. Ήδη λοιπόν ε, βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Θα πρέπει να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του τομέα της άμυνας κάτι με το οποίο βοηθάμε τη χώρα. Πάντως ε, η αφετηρία είναι ήδη πολύ καλή. Ασκήσεις όπως αυτήν που είχαμε τον Ιούλιο, Sea Breeze, με την συνεργασία 19 ε, χωρών του ΝΑΤΟ, όπου είχαμε ε, την αεροπορία, είχαμε επιχειρήσεις στη θάλασσα, ε, αυτές είναι, οι ασκήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ώστε η Ουκρανία να γνωρίζει καλά και την θεωρία και την πρακτική των σύγχρονων επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία επίσης σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλη επιχείρηση του ΝΑΤΟ, Sea Garden, που ξεκίνησε το 2016 στην Ουκρανία και αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται ε, στην οικοδόμηση δυναμικού για την ε, ασφάλεια στη θάλασσα, ε, ευιστοποίηση και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτό δεν είναι κάτι νέο για την Ουκρανία, διότι ήταν μία από τις χώρες που συμμετείχαν στην προηγούμενη επιχείρηση, πριν το Sea Garden, Axe Και συμμετείχε η Ουκρανία με μια φρεγάτα Πολύ σημαντική συμμετοχή. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε με την Ουκρανία για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σε συνεργασία με ε, το Κυβερνείο Θαλασσίων Επιχειρήσεων στην Οδυσσό. Επίσης, είχαμε κάποιες συναντήσεις στην Οδυσσό, κάποιες ασκήσεις που αποτέλεσαν ευκαιρία να αυξήσουμε την ετοιμότητα των ε, ναυτικών δυνάμεων της Ουκρανίας. Επίσης, σε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις του ΝΑΤΟ συμμετέχει η Ουκρανία. Σημαντικό παράδειγμα ήταν Η παρατήρηση ε, στην σημαντική άσκηση Dynamic Mercy στην Δανία και επίσης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην ιατρική διάσκεψη στο Μπέργεν ε, της Νορβηγίας τον Απρίλιο. Συνεργαζόμαστε για να αναπτύξει η Ουκρανία δυνατότητες κατάρτισης δικές της και γενικά στα, στους διάφορους φορείς εντός ε, της άμυνας αλλά και εκτός ε, προσπαθούμε να στηρίξουμε την Ουκρανία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία το 2015. Στηρίζουμε λοιπόν έμπρακτα την Ουκρανία. Αποτελεί σημαντικό τμήμα της καθημερινής μας εργασίας αυτό και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, αλλά και μέσα από μια σειρά εργαλείων του ΝΑΤΟ βοηθάμε την Ουκρανία να πετύχει το στόχο της προσχώρησης στο ΝΑΤΟ. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και κάποια συγκεκριμένα θεσμικά μέσα. Η ιδιαιτερότητα της Ουκρανίας ε, είναι η σχετική επιτροπή με την οποία έχουμε κανονίσει η συνάντηση την επόμενη εβδομάδα ε, για να αξιολογήσουμε την κατάσταση στη θάλασσα του Αζόφ. Ε, θα συναντηθούμε με τον Υπουργό που είναι αρμόδιο ε, για τα κατεχόμενα εδάφη και θα συναντηθούμε και με τον Υπουργό Κλίνκεν πριν από τη συνάντηση αυτή. Κλείνοντας, θα πω ότι είναι σημαντικό για μας να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη Ρωσία όσον αφορά τη συμπεριφορά της απέναντι στην Ουκρανία διότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο προκλητική και στη θάλασσα του Αζόφ. Όπως ίσως γνωρίζετε, συνεχίζουμε να έχουμε συναντήσεις με τη Ρωσία στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας και πάντα η Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή του θεματολογίου μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διαβουλευόμαστε και με την Ουκρανία για να μεταφέρουμε στη Ρωσία μηνύματα σημαντικά για την Ουκρανία, πέρα από τα δικά μας μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις ανησυχίες μας σχετικά με τις συνέπειες των πράξεων της Ρωσίας. Θα έχουμε λοιπόν άλλη μία συνάντηση με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία, όπου θα μπορέσουμε να θίξουμε θέματα όπως είναι η θάλασσα του Αζόφ. Θα κλείσω εδώ. Πολύ ευχαριστώ, Θα προχωρήσω σε περαιτέρω λεπτομέρειες είτε όσον αφορά τις ναι. δικές μας αποτρεπτικές ενέργειες, είτε όσον αφορά την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία που παραμένει πάντα στην κορυφή του θεματολογίου μας. Μια τελευταία παρατήρηση πριν κλείσω. Έχουμε φυσικά και άλλους δύο εταίρους στον Εύξηνο Πόντο, την Γεωργία και τη Μολδαβία, με τους οποίους επίσης έχουμε στενή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άρχεται η συζήτηση, συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Να είστε σύντομοι λοιπόν παρακαλώ. Έχουμε συνεχή επαφή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μέσω του ε, ΠΑΚ που μας επιτρέπει αυτή την συνεργασία συνεχώς με το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου τη Ουκρανική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα και ειδικότερα εσά, κυρία Πρόεδρε, που ε, διατηρείτε την Ουκρανία σε τόσο μεγάλη προτεραιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ του ομιλητέ για τι παρουσιάσει και τι απόψει του για την ε, επιδεινούμενη κατάσταση ε, στη θάλασσα του Αζόφ. Όπως γνωρίζετε, η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας ε, ε, παρακολουθεί με πολύ προσοχή την κατάσταση στην θάλασσα του Αζόφ και γύρω από αυτήν και στην τελευταία συζήτηση του κοινού, της κοινή μας συνεδρίασης με τη Βιχόβνα Ράντα που είναι το κοινοβούλιο του, ε, της Ουκρανίας εκφράσαμε την κοινή μας ε, σύσταση και δήλωση βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην Ανατολική Ουκρανία με την αυξημένη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας και το μπλοκάρισμα των πλοίων ε, μετά ε, την, με την κατασκευή της γέφυρας στο στενό του Κέρτς. Επίσης, ε, όσον αφορά την λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή έχουν συμπεριληφθεί ε, στον κατάλογο των εταιριών ε, με κυρώσεις. Η κατάσταση στη θάλασσα του Αζόφ ε, δεν είναι τόσο πολύ, δεν καλύπτεται τόσο πολύ από τα μέσα ενημέρωσης και είναι δύσκολο να γίνουν δημόσιες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, για μας το πιο σημαντικό ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και πώς μπορεί να βοηθήσει το διεθνές δίκαιο. Εγώ λοιπόν θα ήμουν πάρα πολύ ευγνώμων αν μπορούσαμε να έχουμε πιο λεπτομερείς διευκρινήσεις από τους ομιλητές, πώς θα μπορούσε να είναι επιλογή, να υπάρχει μία αποστολή ανθρωπιστική, ε, ειρηνευτική στην περιοχή από τον ΟΗΕ και ποια θα ήταν η εναλλακτική επιλογή, όπως για παράδειγμα ενδεχόμενη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Θα με ενδιαφέρει επίσης να ακούσω την άποψη του κυρίου Ντεβίνια σε σχέση με τις ε, προτάσεις ε, του κυρίου Γελισέιεφ για περαιτέρω δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κελάμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για τις ε, ομιλίες σας και την παρουσίαση της κατάστασης ε, στη θάλασσα του Αζόφ και στη γύρω περιοχή. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικό γιατί είναι μία σταδιακή προσπάθεια των ρωσικών αρχών να επεκτείνουν την επιρροή τους στη θάλασσα του Αζόφ και αυτό που πρέπει να κάνουμε, συμφωνούμε με τον, συμφωνώ με τον πρέσβη Γελισέγεφ, ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ε, του ομίλου G7 να, να επανεπιβεβαιώσουμε την κυριαρχία της Ουκρανίας ε, στην ε, στο στενό του Κέρτς και αν υπάρξει κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά προφανώς ε, μας απασχολεί το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει σταματήσει δεκάδες εμπορικά πλοία και από την Ουκρανία αλλά και άλλης προελεύσεως, μεταξύ των οποίων ε, και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπό το πρόσχημα των τρομοκρατικών απειλών γίνονται οι επιθερωήσεις στα πλοία αυτά Γι' αυτό λοιπόν αν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να επιβάλλουμε επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Επίσης συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αντιδράσει με πρακτικό τρόπο και να παρουσιάσει νέα επενδυτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των, λιμάνων, των λιμένων ε, Μαριούπολη και Μπερντιάνσκα της ε, Ουκρανίας να βοηθήσει, να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά και ενδεχομένω να παραμείνει η παρουσία των ε, πλοίων ε, του ΝΑΤΟ ε, στον Εύξηνο Πόντο και στη θάλασσα Αζόφ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιούρεκ παρακαλώ έχει το λόγο. Είχατε ζητήσει να λάβετε το λόγο. this. So uh, sorry, I could not follow. I'm sorry, Mrs. Rebecca. Thank you. Κυρία Harms, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση και την παρουσίαση της αποστολής στην Ανατολική Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμμετέχω στη συνεδρίαση γιατί με ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα ε, το, και το πρόβλημα και η λύση του προβλήματος τη κλιμάκωσης θάλασσα του Αζόφ. Γιατί η εντύπωσή μου είναι, και είναι μια εντύπωση που έχουν και άλλοι συνάδελφοι, το ξέρω, το έχω ξανακούσει και πριν από αυτή τη συνεδρίαση, η εντύπωσή μου είναι ότι η αντίδρασή μας δεν είναι καθόλου επαρκής για την ώρα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω κατά πόσο στην ΕΙΕΔ ή στο ΝΑΤΟ υπάρχει συζήτηση για το πώς ακριβώς να αντιδράσουμε και νομίζω ότι είναι ο λόγος νέων τμήματων. Αν δεν υπάρχουν συνέπειες, πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την περαιτέρω επιθετική συμπεριφορά και τακτική της Ρωσίας. Και θα ήθελα επίσης ε, να μάθω αν υπάρχουν συζητήσεις ε, κατόπιν ε, της ε, απόφασης Βαχόφνα Ράντα για το ε, ενδεχόμενο προσχώρησης στο ΝΑΤΟ. Γιατί αυτά είναι τα ζητήματα, τα είναι συνδεδεμένα και δεν μπορούν να παραγνωρίζονται ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ζέμκα, έχετε το λόγο. Θα ήθελα κατερχάς και εγώ να ευχαριστήσω για όλες αυτές τις πληροφορίες, όμως δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνει μόνο όλα αυτά τα οποία ακούσαμε για τη θάλασσα του Αζόφ και επιβεβαιώνει τους φόβους μας. Η Ρωσία δεν θέλει απλώς να διατηρηθεί το status quo, αλλά να επιτύχει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχουν εμπορικά πλοία και πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι αντικείμενο ε, επιθεωρήσεων. Είναι ένας τρόπος πίεσης ε, στην Ουκρανία. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξή. Τι θα κάνουμε. Τρία σημεία θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, να υποστηρίξω οποιαδήποτε δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να βοηθήσει πράγματι την Ουκρανία γιατί έχει όλο το δικαίωμα να περιμένει κάτι τέτοιο η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πιστεύω ότι η κατάσταση σοβαρεύει πολύ και νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά αξιέπαινο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μια κατηγορηματική θέση. Αν λάβουμε μια κατηγορηματική θέση επισήμως θα μπορούσαμε να λάβουμε βρία υποστήριξη. Επίσης, αν δεν απατώμε και αν κάνω λάθος διορθώστε με, η νομική βάση όλων αυτών των επιθεωρήσεων είναι μια, σύμφωνη του 2000, μια συμφωνία του 2003 μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία το χρησιμοποιεί αυτό ως μέσο πίεσης. Είναι όμως ίση εταίροι και συμβαλόμενα μέρη σε αυτήν την συμφωνία. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η Ουκρανία έχει νομικό τη δυνατότητα να κάνει και εκείνη επιθεωρήσεις στα ρωσικά πλοία. Γιατί η Ρωσία αντιδρά στα γεγονότα. Οπότε ίσως θα ήταν ένας τρόπος να δείξει και η Ουκρανία ότι όντως προσπαθεί να αντισταθεί αξίζει τον κόπο. Κύριε Γιούρεκ, ναι, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα το θέμα αυτό. Κύριε Υπουργέ, τι κάνει η Ουκρανία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί είναι μια πλατφόρμα που η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις, ειδικότερα όσον αφορά την Κρυμαία. Ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα αξιολογούσατε τη συμφωνία Μίνσκ σήμερα. Εγγυάται όντως την ειρήνη και την ασφάλεια, ειδικότερα στην Ανατολική Ουκρανία που είναι διαφορετικό από αυτό το πρόβλημα της ε, θάλασσας του Αζόφ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Ζέμκα. Αυτή η διμερή συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της αποστολής μας. Υπεγράφει το 2003 από τις Ουκρανικές ε, αρχές υπό τον πρόεδρο Κούτσμα και από τη Ρωσία. Υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα με την αξιολόγηση αυτής της κατάστασης. Σήμερα όχι μόνο λόγω της παράνομης κατά τη γνώμη μου προσάρτησης της Κρυμαίας, ε, είναι απολύτως σαφές από το 2007 και ειδικότερα και μετά τα γεγονότα στη Γεωργία, την ε, επιθετική πολιτική για τον πόλεμο με τη Ρωσία, Υπάρχει ιστορικά η βούληση, η προσπάθεια να διατηρηθούν ε, κάποιες λεκάνες ε, ή κάποιες θάλασσες όπως ε, του Αζόφ, όπως ο Εύξηνος Πόντος, υπό επιρροή. Το έχουμε δει αυτό και στη Βαλτική θάλασσα. Να είναι δηλαδή εσωτερικές λιμνοθάλασσες και να δημιουργείται έτσι ένα νομικό, στρατιωτικό περιβάλλον, ενδεχομένως και νομικό περιβάλλον. Για να μην υπάρχει πρόσβαση για άλλους εταίρους ή να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι περίπου όμοιο με αυτό του κυρίου Ζβιεύκα. Ε, Τι αντίμετρα μπορεί να υπάρξουν Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάποιοι πυρογνώμονε και μάλιστα προσφάτως το άκουσα κατά τη διάρκεια σε μία συζήτηση πισή στην οποία συμμετείχα. Για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξουν ε, νιοπομπές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ή να βοηθήσουμε στην επιλύση του προβλήματος. Ο κύριος Ντεβίνη πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για, το, για τα ερωτήματα, τους ε, αξιότιμους ευρωβουλευτές. Προφανώς η κατάσταση στη θάλασσα του Άζοφ και οι, κατα... για την ε, ουκρανική ε, οικονομία είναι ένα από τα προβλήματα που προκαλεί η Ρωσία στην Ουκρανία αλλά ήδη γνωρίζουμε αρκετά να μην ξεχνάμε τα 11 δις ευρώ σε δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά όργανα, να μην ξεχνούμε την υποστήριξη ε, στην Ουκρανία. Είμαστε και από τους μεγαλύτερους δωρητές των αποστολών ΟΑΣΕ στην περιοχή. Την υποστήριξη στις εκλογικές αναμετρήσεις ε, για καλύτερη ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι πολλαπλό στην Ουκρανία και ίσως είναι δύσκολο να απομονώσουμε κάποια στοιχεία του εδώ, σε μία δράση δηλαδή. Όταν πρόκειται ε, για τις κυρώσεις, εντάξει δεν χρειάζεται να σας, εξηγώ, να σας εξηγήσω, ότι τα κράτη-μέλη το αποφασίζουν αυτό, είναι αρμοδιότητά τους, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω εξ ονόματός τους, έτσι είναι τα πράγματα. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν αν θα υπάρξουν νέες κυρώσεις. Να προσθέσω επίσης ότι αν τα κράτη-μέλη επηρεάζονται από τις οικονομικές συνέπειες αυτών των καταχρηστικών επιθεωρήσεων που δεν είναι κάτι καινούριο όσον αφορά τη Ρωσία. Θυμάμαι για παράδειγμα ε, τι γινόταν στα φιλανδικά σύνορα το 2013 πριν από τα γεγονότα στον Ντονμπάς όταν η Ρωσία είπε δημοσίως ότι τώρα θα οργανώσουμε 100% επιθεώρηση των φορτηγών ε, στα σύνορα ε, από το 1% στο 100% καταλαβαίνετε ότι σταματάει το εμπόριο, δεν είναι πια επιθεώρηση. Αν λοιπόν τα κράτη-μέλη υφίστανται τις συνέπειες και ε, ζημία, ε, θα πρέπει να αμφισβητήσουν την νομιμότητα αυτών των επιθεωρήσεων των καταχρηστικών ε, βάσει του άρθρου 5 που εξασφαλίζει την ελευθερία της κυκλοφορίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση όσο ε, και καλυμμένη δράση μπλοκαρίσματος. Υπάρχουν και άλλα που κάνουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ειδικότερα για τις κυρώσεις. Αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση νομίζω ότι ο ρόλος των κρατών μελών και ειδικότερα των επηρεαζομένων κρατών μελών ε, αν θέλουν να κάνουν κάτι, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για την χρήσιμη στήριξη και παρατηρήσεις σας. Μετά από την δήλωση της εκπροσώπου από τον ΝΑΤΟ να σας πω εδώ ότι η Ουκρανία προστατεύει το αριστερό πλευρό του ΝΑΤΟ. Η κατάσταση είναι κάπως ιδιαίτερη, επειδή η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι καλό το ΝΑΤΟ να είναι έτσι πιο γενναίο και να δώσει τουλάχιστον στην Ουκρανία ένα σχέδιο δράσης για προσχώρηση στο ΝΑΤΟ γιατί τηρούμε συγκεκριμένα και τα κριτήρια όπως συμβολή ας πούμε στην ασφαλεία περιοχής ε, φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό κλπ. Οπότε είναι ώρα πια να μιλήσουμε για την προσχώρηση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ευχαριστώ την Ριμπέκα Χάρμ που μας υπεθύμησε την πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας να βάλουμε στο Σύνταγμα αυτό το στρατηγικό στόχο για την Ουκρανία, δηλαδή πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Μιλάμε εδώ για τις αξίες και για την βούληση της Ουκρανίας να είναι κοντά στην Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η λογική φυσική μας επιλογή και θα ήθελα να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ επιτυχή διαδικασία στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο για να υιοθετήσουμε τροπολογίες στις αρχές του επόμενου έτους τροπολογίες που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Δικαστήριο για να κάνουμε αυτή ακριβώς την συνταγματική μεταρρύθμιση και αναζητούμε αυτή τη στιγμή τι ε, πλειοψηφίε. Για τον Μπέρκα και τη Μαριούπολη είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούν στενά οι Ουκρανικές αρχές και ο πρόεδρος μάλιστα ιδιαίτερα. Και να σας ενημερώσω ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο πρόεδρος Ουκρανίας θα επισκεφθεί τη Μαριούπολη. Και βεβαίω θα συζητήσουμε το θέμα της αποκατάστασης της περιοχής και το πώς θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε στην επιθετική ρωσική στάση. Πριν ε, λίγες μέρες ο πρόεδρος συγκάλεσε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας που εξέτασε τις ενδεχόμενες αντιδράσεις στην επιθετική στάση της Ρωσίας. Και να τονίσω για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό με διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Κάποιοι από τους προλαλήσαντες μίλησαν για διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας το 2003 στη θάλασσα του Ροζόφ. Αυτό είναι αλήθεια. Και σύμφωνα με αυτή την συμφωνία η θάλασσα αυτή είχε αναγνωριστεί ως εσωτερική θάλασσα και για τη Ρωσία αλλά και για τη Ρωσική Μοσπονδία και για την Ουκρανία. Δυστυχώς όμως οι βασικές η βασική αρχή της συμφωνίας είναι η ελεύθερη διέλευση. Η Ρωσία τώρα καταχράται αυτή της ελεύθερης διέλευσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όλα τα εμπορικά πλοία έχουν νόμιμα δικαιώματα να φέρουν εις πέρα στις εμπορικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ουκρανικούς λιμένες. Η Ρωσία προσπαθεί να τα μπλοκάρει βέβαια όλα αυτά, να τα παρεμποδίσει και αυτό μας προκαλεί σοβαρές οικονομικές απώλειες. Αυτό είναι ένα ζήτημα προβληματικό και μεγάλη πρόκληση για μας. Παραδείγματος χάρη, λόγω αυτού του γεγονότος, ο φόρτος εργασίας μειώθηκε στα ουκρανικά λιμάνια της θάλασσας του Αζόφ κατά 43% λόγω της τάσης της Ρωσίας. Η Ρωσία κάνει ελέγχους επιθεωρήσεις στα εμπορικά πλοία που κρατάνε μέχρι και 6 μέρες, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Επίσης, ξαναλέω, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επόμενες συνεδριάσεις της θα κάνει ξεκάθαρες δηλώσεις για την κατάσταση στην θάλασσα του Αζόφ και την ρωσική επιθετικότητα. Έχουμε το επόμενο Συμβούλιο τον Οκτώβρη, την επόμενη εβδομάδα, οπότε ελπίζουμε αυτή η συνάντηση να συζητήσει αυτό το ζήτημα, να συζητηθεί εκεί και να προχωρήσουμε παραπέρα. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ξέρω ότι και άλλοι είναι ενεργοί στον Τόνμπασκ που θα μπορούσαν βέβαια να εποπτεύουν και άλλοι οργανισμοί που θα μπορούσαν να εποπτεύουν την κατάσταση στα στενά και στη θάλασσα του Αζόφ. Γιατί όχι. Εδώ είμαστε ακριβώς για να συνεργαστούμε ώστε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Και επίσης, το ανέφερε και ο Λουκ, θα βοηθούσε να είχαμε ένα είδο βοήθεια ή αρρωγή. Και να σα το πω ειλικρινά. Βοήθεια που παρέχει αυτή τη στιγμή η Ένωση στην Ουκρανία, αλλά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη η βοήθεια αυτή. Έχουμε την μακροοικονομική βοήθεια προς την ε, Ουκρανία, τουλάχιστον η πρώτη δόση θα έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τα τέλη του μήνα, γιατί για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η Ουκρανία εφαρμόζει τις κύριες παραμέτρους του Μνημονίου Συνεργασίας και γι' αυτό ακριβώς κάνω έκκληση στους φίλους από την Ευρωβουλή να πιέσουν την Κομισιόν ώστε τελικά να ελοπίσει την υπόσχεσή της και να δώσει την πρώτη δόση 500 εκατομμυρίων ευρώ μικρο, μακροοικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα προς όλους και προς τη Ρωσία ότι συμπαραστέκεται στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι και για την ερώτηση για την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι γύρω στο 70% του χρόνου μου στο γραφείο. Να σας πω ότι η Ουκρανία έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει όλες τις υποχρεώσεις της υπό την Συμφωνία του Μίνσκ. Και ένα ζωντανό παράδειγμα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο, στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Πρόεδρου μας για την επέκταση του καθεστώτος, του ιδιαίτερου καθεστώτος, μέχρι το Δεκέμβριο του 2019. Αυτές είναι λοιπόν απτές αποδείξεις της βούλησης των κανονικών αρχών και του Πρόεδρου μας. Δυστυχώς η Ρωσία δεν έχει εφαρμόσει ούτε ένα σημείο από την Συμφωνία του Μίσκ για την ασφάλεια. Γιατί το κύριο θέμα εδώ είναι η ασφάλεια. Δηλαδή, να σταματήσουμε τους θανάτους και τις δολοφονίες των Ουκρανών, να φύγουν τα στρατεύματα τα ρωσικά και να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι, οι κρατούμενοι στις κατεχόμενες περιοχές ώστε να σταματήσουμε τις επιθέσεις προς τις ναυτικές δυνάμεις και να καταστήσουμε καθεστώς ασφάλειας. Ακόμα και το ντίζελ, το καύσιμο, παρακρατούν οι Ρώσοι, ώστε να μην φτάσει στα ρωσικά τάγκς. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο κατεχόμενο των Μπάσκ συζητάμε την εγκατάσταση ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ που θα μπορούσαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη την περιοχή, ακόμα και αυτοί που έχουν γρώσει. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Όταν σταματήσουμε την παρίσφρηση ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού και οπλισμού στην περιοχή, τότε αμέσως θα διευκολύνουμε και θα συμβάλλουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκι για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στο κατεχόμενο Τόνμπασκ. Γι' αυτό ακριβώς Χαίρομαι για την θέση της Γαλλίας και τον ΗΠΑ, ώστε να έχουμε κοινέ θέσει διεθνώ για αυτές τις επιχειρήσεις. Και υπάρχει μόνο μία χώρα η οποία αρνείται να μας στηρίξει. Και ξέρετε ποια χώρα εννοώ. Οπότε, ε, φίλοι, το λέω λίγο συναισθηματικά αυτό, αλλά είναι εύκολο να τελειώσουμε, να θέσουμε τέλος σε αυτή την σύγκρουση σε αυτόν τον πόλεμο. Χρειάζεται μόνο μια πρωτεύουσα να το αποφασίσει και να πιστεί. Γι' αυτό το πρόβλημα δεν είναι η συμφωνία του Μίνσκ, είναι η έλλειψη πολιτική βούληση, επειδή η Ρωσία δεν χρειάζεται το Ντόν μόνο, χρειάζεται ολόκληρη την Ουκρανία. Θέλουν να εφαρμόσουν αυτή τη νέα πολιτική. Γι' αυτό ακριβώ λοιπόν, χρησιμοποιώντα αυτό το υψηλό επίπεδο βήμα, κάνω μια έκκληση να είναι ενωμένη, να μην επιτρέψει στην Ρωσία να μας διασπάσει. Ξέρετε για ποια χώρα μιλάω και ελπίζω τον Δεκέμβρη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει πολιτική απόφαση όχι μόνο για την παράταση των οικονομικών κυρώσεων αλλά για την αύξηση μάλιστα των κυρώσεων αυτών. Γιατί το τίμημα για τη Ρωσία θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά. Αναλογικά με την επιθετική του στάση. Πόσοι Ουκρανοί θα πεθάνουν όταν θα έχουν πεθάνει όταν η, η διεθνής κοινότητα θα πώς θα πεθαίνουν ενώ η διεθνής θα φιλιέται με τους Ρώσους ηθήνοντες σε αυτές τις εκδηλώσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση. Θα ήθελα λοιπόν να ξανατονίσω την ηγετική στάση Μέρκελ και Μακρόν εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βελισεύ. Η κυρία Στεφανόβα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε κυρία Στεφανόβα παρακαλώ γρήγορα. Θα αναφέρω πολύ σύντομα τέσσερα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ερώτηση και σας ευχαριστώ για την πολύ εύστοχη αυτή ερώτηση σχετικά με το ΝΑΤΟ και την ε, κατάσταση ασφαλείας ε, στη θάλασσα του Αζόφ. Ναι, όπως ανέφερα στην παρουσίασή μου, όχι μόνο παρακολουθούμε ε, στενά την κατάσταση, αλλά και στο στρατηγείο στις Βρυξέλλες ε, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και με την Ουκρανία και την Γεωργία έχουμε σχετική συνεργασία. Είπαμε ότι η προσάρτηση της ε, Κρυμαίας υπονομεύει την ε, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή ε, και η οικοδόμηση της γέφυρας στο στενό του Κέρτς επίσης αποτελεί προκλητική ενέργεια. Το έχουμε πει αυτό, λοιπόν, το έχουμε καταδικάσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο Γενικός Γραμματέας Στόλτενπερκ το ανέφερε αυτό σε σχετική διάσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα που μίλησε για τα εμπόδια στην εμπορική ναυτιλία και αυτό με φέρνει στο δεύτερο θέμα που ήθελα να αναφέρω. Τι να κάνουμε. Δεν θα σχολιάσω τις κυρώσεις, αυτό είναι θέμα που θα πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από πλευράς του ΝΑΤΟ πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά ε, τι κάνουμε. Αλλά για να αποτρέψουμε την Ρωσία θα πρέπει να ε, λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ε, το κάνουμε αυτό, για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία θα θίξουμε το θέμα της θάλασσας στο Αζόφ. Είναι σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Πρέσβης, είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό από όλες τις πλευράς, διότι δεν διαφωνούμε όσον αφορά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η παράνομη κατασκευή της γέφυρας και η κατάσταση στη θάλασσα του Αζόφ σίγουρα αποτελούν κλιμάκωση όσον αφορά την κατάσταση ασφαλείας. Επίσης είχαμε το θέμα των συνταγματικών τροποποιήσεων ώστε να συμπεριληφθεί η ε, συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σύνταγμα της ε, Ουκρανίας. Ε, ναι, παρακολουθούμε στενά και το θέμα αυτό, το συζητάμε με τους Ουκρανούς ε, εταίρους μας. Βέβαια, το θέμα του συντάγματος είναι θέμα της Ουκρανίας. Όσον αφορά την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ, η ηγεσία του ΝΑΤΟ αναγνώρισε τις προσδοκίες της Ουκρανίας για προσχώρηση. Αυτό δεν είναι κάτι νέο, αυτό ξεκίνησε το 2008 που λάβαμε απόφαση και η πόρτα του ΝΑΤΟ παραμένει ανοιχτή. όπως ήδη φάνηκε με την προσχώρηση του Μαυροβουνίου πέρσι και την έναρξη των συνομιλιών με την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας φέτος. Ο φίλος μου και πρέσβης ε, γνωρίζει πολύ καλά ότι είχαμε επανειλημμένα τη συζήτηση αυτή και μεταξύ μας ε, και με άλλους ε, Ουκρανούς συναδέρφους. Η Ουκρανία έχει σημειώσει εκπληκτική πρόοδο, ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ακόμα περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια. Συνεργαζόμαστε στενά, όπως σας είπα, για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να ε, φτάσει να πληρεί τις προϋποθέσεις για προσχώρηση και απομένουν κάποια πράγματα που πρέπει ακόμη να ε, έχετε, όπως για παράδειγμα η δημοκρατική πολιτική, ε, ο δημοκρατικός πολιτικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το στόχο σας, το αν θα γίνει αυτό μέσω του, μέσω του συντάγματος ή μέσω άλλου τρόπου, αυτό εναπόκειται σε εσάς. Και μία τελευταία παρατήρηση, διότι καταλαβαίνω ότι καθυστερήσαμε. Η νομική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην Ουκρανία έχουμε μια πολύ ζωντανή εσωτερική συζήτηση σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της εγκατάλειψης ε, της συνθήκης του 2003 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ε, σχετικά με τη χρήση της θάλασσας του Αζόφ. Διότι ε, πάντα με εντυπωσίαζε στην Ουκρανία η ζωντανή κοινωνία των πολιτών. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή. Εναπόκειται στην Ουκρανία να λύσει το θέμα, αλλά είχαμε πρόσφατα μελέτη, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε μελέτη για το θέμα αυτό που παρουσιάζει το θέμα πολύ ολοκληρωμένα. Θα στηρίξουμε λοιπόν αυτά που κάνει ήδη η Ουκρανία, δηλαδή να προσπαθήσει να λύσει τα θέματα αυτά με διπλωματικά και νόμιμα μέσα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, πρέπει να κλείσουμε το θέμα αυτό της συζήτησης. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας. Σας παρακαλώ να τους χειροκροτήσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ε, έρθουν στο βήμα, θα έρθει στο βήμα ο επόμενος ομιλητής και θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε. Πολύ λυπάμαι για την καθυστέρηση. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης, που είναι η παρουσίαση της μελέτης με θέμα την τυποποίηση του ευρωπαϊκού εξοπλισμού. και θα ήθελα να προσκαλέσω, να καλωσορίσω τον κύριο Ντάνιελ Φιότ που είναι εμπειρογνώμων του EUISS, του Ινστιτούτου Μελετών για Θέματα Ασφαλείας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ την Πρόεδρο. και ευχαριστώ και το τμήμα ε, μελετών που μας ανέθεσε τη μελέτη αυτή. Ήταν ε, τιμή και προνόμιο για μας να αναλάβουμε αυτήν την μελέτη. Παρότι είναι ιδιαίτερα τεχνικό το θέμα, θα πρέπει να σας πω ότι πέρασα πολύ καλά γράφοντας τη μελέτη αυτή το καλοκαίρι. Ελπίζω και εσείς να την απολαύσετε εξίσου. Έχουμε εδώ μια παρουσίαση στις οθόνες. I can control it. I have full control over the uh, presentation. Ωραία, έχω τον απόλυτο έλεγχο της παρουσίασης. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε τους στόχους της μελέτης γενικά. Τι ζητήθηκε δηλαδή από μένα και το Ινστιτούτο EU Πόσο αποτελεσματικές ε, ήταν οι προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τυποποίηση του εξοπλισμού μέχρι τώρα και όσον αφορά το μέλλον, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι προσπάθειες αυτές και να ε, επεκταθούν και σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς πολιτικής. Ιδιαίτερα μου ζητήθηκε να επικεντρωθώ στο θέμα της ανταλλαγής ε, πληροφοριών στη θάλασσα και το άπχας, δηλαδή συστήματα πιλωτικά εξαποστάσεως. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς μπορεί να ε, επεκταθεί η τυποποίηση και σε άλλους τομείς. Γενικά η μελέτη εξετάζει πώς η επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού μπορεί να πάει στο μέλλον και επίσης είχαμε και μια δευτερεύουσα ερώτηση σχετικά με την σύγκριση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όσον αφορά την τυποποίηση. Φυσικά το πρώτο τμήμα οποιασδήποτε μελέτης ε, είναι να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογή ε, της μελέτης. Ε, η τυποποίηση της άμυνας, η τυποποίηση του εξοπλισμού είναι ένα θέμα ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν είναι πάντα όμοια τα στρατιωτικά συστήματα τυποποίησης με τα πολιτικά. Αλλά ο γενικός στόχος της τυποποίησης φαίνεται εδώ στη διαφάνεια είναι η διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενη ε, χρήση κατευθυντηρίων γραμμών ε, για να ε, έχουμε τις ίδιες διαδικασίες και κανόνες. Δηλαδή, εάν εντοπίσουμε και κατηγοριοποιήσουμε και εάν παρέχουμε ακόμη στοιχεία για τα διάφορα συστήματα, οι διαδικασίες θα είναι πολύ πιο απλές, αποτελεσματικές και θα αποφύγουμε τον κίνδυνο επικάλυψης εργασιών και ε, κόστους. Άλλο σημαντικό στοιχείο κλειδί στον ορισμό της τυποποίησης, ιδιαίτερα όσον αφορά την τυποποίηση στον τομέα της άμυνας, είναι η διαλειτουργικότητα. Ο στόχος ε, της τυποποίησης των στοιχείων και τεχνολογιών είναι ότι θεωρητικά τουλάχιστον τελικά τα συστήματα άμυνας θα είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους και εντός της ίδιας χώρας, ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες και μεταξύ χωρών. Δηλαδή, είτε αυτό είναι στο πλαίσιο της ΕΚΕΠΑ, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Επίσης, κάτι ακόμα θα πρέπει να έχουμε κατά νου κατά τη συζήτηση τη τυποποίηση, τη διαφορά ανάμεσα στην τυποποίηση στην άμυνα και την πιστοποίηση ή τον καθορισμό ε, κοινών απαιτήσεων για τις ε, δυνατότητες που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Η τυποποίηση γενικά αναφέρεται σε στοιχεία και τεχνολογίες, ενώ η πιστοποίηση, όπως και οι εναρμονισμένες κοινέ απαιτήσει, ε, έχουν να κάνουν με συμφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τον βιομηχανικό τομέα ή με τις ένοπλες δυνάμεις ότι θα ε, υπάρξουν κοινέ προδιαγραφές για ό,τι σύστημα άμυνας θέλουν να αναπτύξουν. Δηλαδή, αν έχουμε μια κοινή συμφωνία μεταξύ κρατών μελών ότι από κοινού θα αναπτύξουν ένα σύστημα άμυνας ή ένα συγκεκριμένο κομμάτι τεχνολογίας, αυτό θα αυξήσει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας και θα μειώσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την επικάλυψη εργασιών και το κόστος. Επίσης ε, σημαντικό είναι το, να έχουμε κατά νου το γενικότερο πλαίσιο της τυποποίησης ε, στην άμυνα. Κάτι που είναι προφανές από κάθε μελέτη είναι ε, η ασαφής διακριτική γραμμή ανάμεσα στον πολιτικό και τον στρατιωτικό τομέα. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της συζήτησης. Όλο και περισσότερο λοιπόν βλέπουμε ότι κάποια στοιχεία και κάποιες τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα άμυνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, τα πρότυπα αυτά και, τα, και οι τεχνολογίες ε, μπορούν να προέρχονται από τον πολιτικό τομέα. Αυτό λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστου στο να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στον πολιτικό τομέα. Υπάρχει λοιπόν ε, εδώ πέρα μια σαφής διακριτική γραμμή ανάμεσα στους δύο τομείς. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι αυτό, και αυτό σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία, είναι ότι τα πρότυπα είναι εθελοντικά, ούτε καν εντό του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει ένας γενικός μηχανισμός που να ε, επιβάλλει την χρήση προτύπων στα κράτη-μέλη και στους συμμάχους. Ε, η ανάπτυξη των προτύπων είναι κάτι που ξεκινάει από τη βάση και προς τα πάνω. Ε, αυτό ε, αναπτύσσεται στη βιομηχανία ήδη σε πολύ πρώιμο στάδιο και ω μέρος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να υπάρχει συνένεση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν. Αν δεν υπάρχει τέτοια συνένεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο καταρχά να υιοθετηθούν τα πρότυπα και δεύτερον να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα που είναι και ο στόχος της ανάπτυξής τους. Όπως σας είπα, το είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αποφευθεί η επικάλυψη εργασιών και να κρατηθεί χαμηλά το κόστος. Επίσης, σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι παρότι βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικές ανταλλαγές ανάμεσα στον πολιτικό και τον στρατιωτικό τομέα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον καθένα από αυτούς τους δύο τομείς. Και φαίνεται και στη μελέτη ότι για κάποιες τεχνολογίες και για κάποια στοιχεία είναι πολύ διαφορετικές οι απαιτήσει από ε, τον τομέα της άμυνας ε, από ότι η λογική που βοηθάει στην ανάπτυξη προτύπων στο πολιτικό τομέα. Καταρχάς, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι σαφή τα όρια ανάμεσα στους δύο τομείς, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ε, επίσης ο τομέας της άμυνας σε τι βαθμό και σε ποιο στάδιο θα πρέπει να συμμετάσχει στην ανάπτυξη κοινών προτύπων. Αυτό είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, πόσο μάλλον που η ανάπτυξη προτύπων είναι θελοντική από τη φύση της. Υπάρχουν κάποιοι σαφείς τομείς διαφορών για κάποιες τεχνολογίες και στοιχεία. Ε, το επίπεδο ασφάλειας τους είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ε, βλέπουμε στον πολιτικό τομέα. Βλέπουμε λοιπόν προτίμηση για πιο ασφαλή πρότυπα και πιο τεχνικά πρότυπα από ό,τι στον πολιτικό τομέα. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται η διαφάνεια αυτή, αλλά στη μελέτη είναι σαφή τα θέματα αυτά. Ε, πρέπει να γίνουν διάφοροι συμβιβασμοί ε, κατά την τυποποίηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις κοινέ στρατιωτικές απαιτήσει, υπάρχει ε, η σχέση ανάμεσα σε αυτά που καθορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΝΑΤΟ ε, ή τις απαιτήσει ε, σε εθνικό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν την αντίθεση αυτή, την αντίθεση ανάμεσα σε ε, τις κοινέ απαιτήσει και τις εθνικές απαιτήσει. Επίσης έχουμε το θέμα της επικάλυψης ερευνών και τεχνολογιών και των σχετικών δαπανών στα κράτη-μέλη, που φυσικά είναι ε, η λογική του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θέλουμε δηλαδή να ξεφύγουμε από το πρόβλημα αυτό. Κάτι που φαίνεται να είναι και πρόβλημα στον τομέα της τυποποίησης του εξοπλισμού. Τίθεται και το ερώτημα σε ποια φάση της δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να έχουμε τυποποίηση. Ήδη ε, στο στάδιο της τεχνολογικής ετοιμότητας, ε, δηλαδή κατά τη βασική έρευνα, ε, κατά την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή Εάν αναπτυχθούν πρότυπα ε, πιο μετά, ποιο θα είναι το κόστος. Η μελέτη λοιπόν λέει ότι αν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκή συζήτηση για, την, για τα πρότυπα, αυτό θα πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς ε, κατά τη ε, διαδικασία ανάπτυξης, δηλαδή στη φάση ε, έρευνας και τεχνολογίας ή έρευνας και ανάπτυξης. Θα υπάρχει όφελος λοιπόν εάν η τυποποίηση γίνεται όσο γίνεται νωρίτερα και θα πρέπει να έχουμε κατά νου κατά την ανάπτυξη προτύπων ότι αυτό που προσέξαμε σε πολλές ε, δημόσιες συμβάσεις και σε πολλά προγράμματα ε, δημοσίας, ε, δημοσίων προμηθειών προβλήματα ανέκυψαν λόγω της έλλειψης τυποποίησης σε αρχικά στάδια ε, της ε, ε, Σύμβασης Εξοπλισμού. Θα πρέπει λοιπόν οι στρατηγικές τυποποίησεις να εισαχθούν σε πολύ νωρίτερο στάδιο του κύκλου της δημόσιας σύμβασης, της δημόσιας προμήθειας, διότι αλλιώς θα υπάρχει τεράστιο κόστος όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση. Έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε μεγάλο μέρος του κόστους συντήρησης ε, των τεχνολογιών αυτών. Και κάτι ακόμα πρέπει να αναφέρω, την ε, ασφάλεια προμήθειας. Η τυποποίηση είναι ε, σε μεγάλο βαθμό πολιτική διαδικασία, ενώ είναι εθελούσια το να εξεταστεί το τι πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, έχει να κάνει γενικά με την ε, προμήθεια συστημάτων όπλων στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν στην αλυσίδια εφοδιασμού ε, οι διάφοροι παράγοντες να συμμετάσχουν ήδη από την αρχή, διότι πρέπει μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μεσαίου κεφαλαίου να έχουν πρόσβαση στα πρότυπα όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλιώς θα έχουμε κατακαιρματισμό και έτσι η δυνατότητα τυποποίησης και ο εντοπισμός κοινών ε, απαιτήσεων ε, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και πάλι δεν είμαι ε, βεβαίως πόσο σαφής είναι η διαφάνεια, πόσο καθαρή είναι η διαφάνεια, αλλά εδώ βλέπετε πρότυπα που ήδη έχουν αναπτυχθεί ε, στο ευρωπαϊκό τοπίο. Βλέπετε διάφορους ε, παράγοντες, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε το ΝΑΤΟ, που επίσης υιοθετεί πρότυπα. Έχουμε όμως και μια σειρά εθνικών φορέων τυποποίησης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε επίσης φορείς και επιτροπές που είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη ε, προτύπων για τον πολιτικό τομέα. Αλλά στο διάγραμμα αυτό βλέπετε ότι υπάρχει πολύ πιο μεγάλος αριθμός προτύπων για τον πολιτικό τομέα από ότι για τον τομέα ε, Τη άμυνα, διότι είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθούν τέτοια πρότυπα. Ωστόσο, εάν εξετάσετε τους τομείς στους οποίους εκπονούνται τέτοια πρότυπα, ε, για παράδειγμα ε, συστήματα ηλεκτρικής διαλειτουργικότητας, ε, όπως είναι υπολογιστές κλπ. αυτό είναι ένας τομέας που αφορά και τον τομέα της άμυνας. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς λοιπόν ότι Χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο σαφείς όσον αφορά το τι πρότυπα ήδη έχουν αναπτυχθεί στον πολιτικό τομέα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της άμυνας γενικότερα. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Όσον αφορά τις ε, διαφορές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ έχει πολύ πιο μακρά ιστορία εκπόνησης ε, προτύπων πρότυπα υπήρχαν ήδη από την ε, αρχή της συμμαχίας, δηλαδή δεκαετία του 50 και του 60, όπου ήδη υπήρχαν ομάδες εργασίας για την τυποποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρά πείρα ανάπτυξης προτύπων ε, στον ε, πολιτικό τομέα, ενώ δεν φαίνεται να έχει κληρονομιά κατά παράδοση στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα όσον αφορά κάποια στοιχεία προστιθέμενης αξίας ε, που ε, μπορεί να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχά όπως σα είπα, ε, τα όρια ανάμεσα στους δύο τομεί το πολιτικό και το στρατιωτικό, είναι ασαφή. Υπάρχει δυνατότητα υιοθέτηση από τον τομέα άμυνας των όσων έχουν γίνει στον πολιτικό τομέα. Αυτό λοιπόν είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, στοιχεία από τον πολιτικό τομέα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ. Κατόπιν έχουμε το θέμα της νομοθεσίας, διότι υπάρχουν σημαντικά νομοθετικά μέσα που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τις δύο οδηγίες το 2009 ε, για ε, τα, τα, τα συστήματα εξοπλισμού, κάτι που αγγίζει και θέματα τυποποίησης πρέπει να δοθεί πολύ περισσότερη προσοχή στο θέμα της τυποποίησης ε, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής των δύο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άλλος τομέας όπου διαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ΝΑΤΟ, κάτι που θα είναι όλο και πιο σημαντικό στη συζήτηση για την τυποποίηση, έχει να κάνει με ε, τον προϋπολογισμό. Για πρώτη φορά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οικονομικά κίνητρα για να αυξήσει όχι μόνο τον ε, εντοπισμό κοινών απαιτήσεων, αλλά για να χρησιμοποιηθεί η ε, τυποποίηση σε όλους ε, τους τομείς της άμυνας που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Γνωρίζω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ότι παρότι αναφέρονται τακτικά η ανάπτυξη προτύπων και η τυποποίηση, ε, πιο προ... πολύ προτίμηση φαίνεται να δίδεται στην εναρμόνιση των κοινών απαιτήσεων και το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα, αλλά θα ισχυριζόμουν ότι χρειάζεται να εξεταστεί πολύ περισσότερο η τυποποίηση των ε, στοιχείων και τεχνολογιών που κάποια στιγμή θα ενσωματωθούν ε, στις ε, αμυντικές δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ λοιπόν και οι δύο ασχολούνται με την τυποποίηση εξοπλισμού, αλλά έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις και έχουν διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή τους. Ας εξετάσουμε και κάποια υπάρχοντα εργαλεία και πρωτοβουλίες για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί με το θέμα της ε, τυποποίησης στον τομέα της άμυνας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο ε, όσον αφορά την ανάπτυξη σημαντικών βάσεων δεδομένων. Και εδώ στην διαφάνεια βλέπετε ιδιαίτερα δύο το ETSIS και το ETSAR που είναι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων πρόκειται για μητρώα υπαρχόντων προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, από ε, φορείς, ε, κυβερνήσεις κλπ. στον τομέα της άμυνας. Είναι μια ενιαία θηρίδα για αυτούς τους φορείς. Μία από τις ε, συστάσεις μου στην έκθεση είναι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να αντικαταστήσει κανείς ε, ή να καταργήσει αυτές τις βάσεις δεδομένων. Νομίζω ότι εξυπηρετούν... Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά θα μπορούσε να δοθεί πολύ περισσότερη προσοχή Ε, στην ε, κατάργηση προτύπων ε, περιτών. Έχουμε πολλά παλαιότερα πρότυπα, τα οποία μπορεί να ήταν χρήσιμα κάποια στιγμή, δεν έχουν ακολουθήσει όμως τις εξελίξεις στην τεχνολογία και υπάρχουν εκατοντάδες άχρηστα πρότυπα, πεπαλαιωμένα πρότυπα στην αγορά. Στο Έτσι και το Star λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ποια πρότυπα είναι ξεπερασμένα ώστε οι διάφοροι φορείς να γνωρίζουν ποιοι ε, έχουν κατέβει από το ράφι, ποια πρότυπα έχουν καταργηθεί και ποια είναι ακόμη χρήσιμα. Επίσης, έχουμε την ιδέα των υβριδικών προτύπων ε, που σχετίζεται με τα σαφή όρια ανάμεσα στον πολιτικό και τον ε, αμυντικό τομέα. και έχουμε την ε, δημιουργία ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης ε, που έχουν πολύ μεγάλη πείρα στον πολιτικό τομέα και μπορούμε να δούμε τι προστιθέμενη αξία μπορούν να φέρουν στην τοποποίηση του εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στη διαφάνεια αναφέρω τα, τους τρεις βασικούς οργανισμούς ε, όπου βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την Επιτροπή για την ε, τυποποίηση, την Επιτροπή για την τεχνική τυποποίηση και, την, ε, και τον Οργανισμό για την τυποποίηση στις τηλεπικοινωνίες. Μπορούν να βοηθήσουν ε, τον αμυντικό τομέα να εντοπίσει χρήσιμα πρότυπα από τον πολιτικό τομέα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό θα είναι να Πολύ πιο σημαντικό είναι μάλλον ότι συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες ήδη σε πρώιμο στάδιο. Επίσης, σε περισσότερη λεπτομέρεια μπαίνω όσον αφορά την ε, ε, ε, τυποποίηση στον τομέα της ασφάλειας της θάλασσας και των τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων πλοήγησης να σας δείξω που είμαστε σε αυτή τη φάση σε σχέση με την τυποποίηση όσον αφορά την ανταλλαγή ε, ναυτικών ε, ε, πληροφοριών. Υπάρχει ένα δίκτυο για τα δεδομένα των θαλασσών ασφαλές που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό έχει να συμμετέχουν όλες ε, οι ε, αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν καλύτερα να ανταλλάσσουν ε, απόψεις για την περιβαλλοντική προστασία, θαλάσσια δεδομένα, θαλάσσια ασφάλεια κλπ. Για να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ άλλων. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας μας βοήθησε και πάλι τα προγράμματα κατηγορίας Β ή τα προγράμματα ε, ε, παρακολούθησης αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να προσπαθήσουν να αναπτύξουν κατάρτιση μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να εξακολουθούμε να συνδυάζουμε κονδύλια από την ΠΕΣΚΟ ε, και από το Ταμείο Άμυνας ε, και ε, το πρόγραμμα για το 2020 ο ωκεανός 2020 είναι πολύ σημαντικό προσπαθεί να συμπεριλάβει κάποια πιλωτικά προγράμματα στον τομέα των θαλασσών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτύξει το είδος των τεχνολογιών που ε, χρειάζεται για μη επανδρομένα ή τηλεκατευθυνόμενα ε, ε, συστήματα, αλλά είμαστε ακόμη σε ένα πολύ εμβριακό στάδιο. Το πρόγραμμα PESCO το Habsburgo pesco ε, πρόγραμμα που αφορά ε, την ε, θαλάσσια προστασία και παρακολούθηση. Κάποια κράτη-μέλη στο πλαίσιο της Πέσκο το έχουν δρομολογήσει με σκοπό καλύτερη επικοινωνία για τα συστήματα προστασίας των λιμένων και προσπαθήσουν αυτό να το συμπεριλάβουν σε μια ευρύτερη εικόνα της θαλάσσιας προστασίας. Υπήρξαν κάποια κάποιες προσπάθειες, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Στο πρόγραμμα Οκεανός 2020 είναι κάτι που προέκυψε από το πιλωτικό πρόγραμμα. Το ζήτημα είναι πώς αυτό ε, θα συνεχιστεί μετά το 2020 και για το πρόγραμμα ΠΕΣΚΟ είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Τώρα, όσον αφορά τα ε, τηλεκατευθυνόμενα συστήματα αεροσκαφών, κάτι το οποίο ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι η πρωτοβουλία που έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και των αρχών των κρατών μελών το πρόγραμμα ARWA ε, το οποίο σκοπό έχει να συμπεριλάβει κάποια ε, στοιχεία ε, ώστε να μην υπάρχει, μη, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των πληροφοριών στον εναέριο χώρο. Αυτό είναι κάτι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ένα ακόμη υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που ανέπτυξε και προσπαθεί να εξελίξει πρότυπα λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων ε, προκλήσεων στην άμυνα να προσπαθήσει να συμπεριλάβει και ε, τις εμπειρίες τις μη ε, στρατιωτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, γιατί υπάρχουν προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που ε, σκοπό έχει να αναπτύξει διαδικασίες πιστοποίησης και τυποποίησης για τον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο και το πρόγραμμα Τράουα υπό το πιλωτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Ανάπτυξης 455.000 ευρώ περίπου για να υπάρχουν συστήματα ανείχνευσης και για να χρησιμοποιεί ε, ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, αλλά θα συνεχίσω προχωρώ στις συστάσεις, τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επεκτείνει τη δουλειά της και όπως είπα στην αρχή, μίλησα για στρατιωτική κινητικότητα. Μου φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο στο πλαίσιο του ότι η στρατιωτική κινητικότητα είναι πολύ σημαντική και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν μιλάμε για την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο του στρατιωτικού τομέα. Ίσως θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια πρότυπα ε, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε προγράμματα πολιτικά, ε, υποδομές πολιτικές, οι οποίες θα μπορούν να βασιστούν και οι στρατιωτικές κρίσεις. Δεν αφορά μόνο προγράμματα αφορά υποδομές ε, μεταφορών, οδικά, σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια κλπ. Και κάποια συστήματα παρακολούθησης που θα αναπτυχθούν ε, φυσικά στο πλαίσιο των υποδομών μεταφορών. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να παραγνωρίζετε το κομμάτι της τυποποίησης και σε αυτό. Μία ακόμη, ένας ακόμη τομέας που είναι αυτονόητος είναι η κυβερνοασφάλεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα μακρά συζήτηση για το πόσο σημασία έχει η σχέση ε, και η μικρή διακριτή γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στο στρατιωτικό και μη στη στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και στην ΠΕΣΚΟ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας γιατί μπορούν πάρα πολλά προγράμματα να οδηγήσουν στο είδος των ικανοτήτων που θέλουμε να αναπτύξουμε. Κάτι ακόμη, διαχείριση της ενέργειας στον τομέα της άμυνας είναι πάλι ένα πρόγραμμα, ένας τομέας που, στον οποίο επικεντρώνει ο Ευρωπαϊκός οργανισμός άμυνας. Εγώ λέω στην έκθεσή μου ότι πρέπει να δούμε κατά πόσο πολιτικά πρότυπα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί το κόστος διαχείρισης της ενέργειας και του περιβάλλοντος στον τομέα της άμυνας συστάσεις, ε, μία αρκετά ε, χαρακτηριστική και παραδοσιακή, να υπάρχει δηλαδή ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας. Είπα ότι αυτό είναι μάλλον κλισέ, είναι όμως και σημαντικό γιατί ένα από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις μου με τον κλάδο, με την, ε, τον κλάδο της άμυνας είναι ότι εξαιρούνται ε, αποκλείονται από τον τομέα τυποποίηση και ότι θα ήθελα να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία από την αρχή. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση μεταξύ ε, των ε, αμυντικών εταιριών και των ε, ε, πολιτικών εταιριών ε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια ομάδα επαφής για την τυποποίηση στην άμυνα, για να μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ο αμυντικό τομέα νωρίτερα στη διαδικασία. Δεν λέω ότι δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου. Αν δούμε λίγο, λίγη από τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα, το, το διαπιστώνουμε. Αλλά όταν βλέπει κανείς από πιο μακριά τα πράγματα, βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στον, στην ανάπτυξη προτύπων, ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη σχέση με τους ε, φορείς, ε, τους μη στρατιωτικούς και του τομέα της άμυνας. Το δεύτερο όμως συμπέρασμα είναι βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει μία μόχλευση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει τώρα, ε, να υπάρχει τυποποίηση ε, στον τομέα της άμυνας, όχι γιατί υπάρχει μόνο το πρόβλημα των οικονομικών κινήτρων, δηλαδή δυνατότητα να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να ενθαρρύνουμε περισσότερη τυποποίηση πέρα από την παραδοσιακή εθελοντική συμμετοχή, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το Ταμείο Άμυνα, γιατί αν δεν υπάρχει τυποποίηση από τα αρχικά στάδια, τότε τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Άμυνα μπορεί να ε, χαρακτηρίζονται από τα ίδια προβλήματα που είδαμε σε προ... πολυμερή προγράμματα συνεργασία εκτό του Ταμείου. Δεν υπάρχουν κοινέ απαιτήσει, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα, δεν υπάρχει διαχείριση του κόστου που έχουν κάνουν με την απόδοση, όλα αυτά προκύπτουν από τη μη τυποποίηση. Ε, αν δεν υπάρχει τυποποίηση, αν δεν γίνει σωστά η τυποποίηση, μπορεί να, υπάρχει, να υπάρχουν προβλήματα και στο πλαίσιο του Ταμείου Άμυνα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να τα αποφύγουμε. όσον αφορά τώρα το ΠΕΣΚΟ, Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξη ικανοτήτων και στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ, εναρμόνιση απαιτήσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα προγράμματα υπό τον ΠΕΣΚΟ ε, και αυτό το λέω κυρίως εν ώψη για της περίοδου μετά το 2020 κυρίως. Αυτά τα προγράμματα που αναπτύσσονται εντός της ΠΕΣΚΟ αλλά και με τη χρήση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, αν λοιπόν αυτά τα προγράμματα μεταξύ των δύο φορέων που αναπτύσσονται και από τους, μεταξύ των δύο φορέων και από τους δύο φορείς, το ερώτημα είναι πώς θα γίνει η διαχείριση της τυποποίησης σε ένα πλαίσιο που έχουμε από τη μία την ΠΕΣΚΟ που ξέρουμε ότι είναι ε, σε μεγάλο βαθμό διακυβερνητική και από την άλλη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που, παίρνει, έχει ένα χαρακτήρα πολύ πιο υπερεθνικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο συνοχή γιατί θα έχουμε το Ταμείο της Άμυνας και θα έχουμε και την ΠΕΣΚΟ και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την τυποποίηση. Τέταρτον, να προσπαθήσουμε περισσότερο να ενσωματώσουμε το κομμάτι της τυποποίησης στα νομοθετικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα λόγω της οδηγίας ε, για, μεταφο για τις με για μεταφορών, το θέμα της αλυσίδας εφοδιασμού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πλέον στον τομέα της άμυνας και το, και το βλέπουμε αυτό και λόγω της άφηξης της ΠΕΣΚΟ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Κάθε φορά που υπάρχει νομοθεσία, ως μήμα της διαδικασίας αξιολόγησης θα πρότεινα ένα από τα σημεία της ε, διαδικασίας να είναι πόσο έχουμε προχωρήσει στον τομέα της τυποποίηση. Και θα έλεγα ότι είναι ένα ευρύτερο ζήτημα αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουμε βάσεις δεδομένων, ομάδες επαφών με, που, προ, που προβαίνουν στην τυποποίηση άμυνας, δεν έχουμε τρόπο να αξιολογήσουμε πόσο επιτυχής ήταν αυτή η διαδικασία τυποποίησης και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το σκεφτούμε περισσότερο. Και τέλος και θα ολοκληρώσω, για να μην επαναλαμβάνομαι συνεχώς, είναι η βελτιστοποίηση των βάσεων δεδομένων και των μητρών που έχουμε. Δεν είναι μόνο ένα θέμα που αφορά ότι υπάρχει, το ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια, κάποιος βαθμός συνοχής μεταξύ ε, των ε, μητρών του ΝΑΤΟ αλλά ε, τα θέματα του κατά πόσο κάποια συστήματα είναι παροχημένα, ε, να δούμε δηλαδή ε, τι πρότυπα μπορεί να χρειαζόμαστε και για το μέλλον, να τα εντοπίσουμε. Όλα αυτά μπορούν να παίξουν πάρα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο στο να προσπαθήσει να προβλέψει ο τομέας τι πρότυπα θα χρησιμοποιούνται σε ένα τοπίο που συνεχώς αλλάζει. Και εδώ κλείνω την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή σας παρουσίαση και την πολύ καλή σας έκθεση. Το ερώτημά μου είναι κάποια πεπαλαιωμένα πρότυπα. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα εκπνοής χρειαζόμαστε μία ad hoc προσέγγιση και μία ρεαλιστική προσέγγιση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών ε, οργάνων. Για τη στρατιωτική κινητικότητα. Φαίνεται ότι στις αρχές των επιχειρήσεων ε, του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ήταν μία προϋπόθεση της, της κινητικότητας, η υποδομή δηλαδή, να εξασφαλίζεται κάποια τυποποίηση για να εξασφαλίζεται και η κινητικότητα. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό τώρα. να το, να το εισαγάγουμε αυτό στο τρέχον πι ή στο επόμενο. Τι χρειαζόμαστε ακριβώς. Uh, next uh, with the... Τι χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας μεταξύ άλλων εδώ στην υποεπιτροπή μας τονίσαμε το ρόλο, το, τη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου του Ταμείου αυτού. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να, να, ε, να κάνουμε για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε και από τη διαδικασία της τυποποίησης. Uh, thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι μια μη επιτυχημένη, μακρά η ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια. Ε, δεν είχαμε κανένα απτό αποτέλεσμα. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε νέες πολιτικές, αναφερθήκατε σε κάποιες από αυτές και το ερώτημά μου είναι σε σχέση με την ανάπτυξη υποδομών, το σχετικό πρόγραμμα και την ε, ετήσια έκθεση ε, που αφορά την άμυνα. Πώς μπορεί αυτές οι δύο πολιτικές να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σημαντικότερα βήματα προς την τυποποίηση. Κύριε Γιούρεκ, έχετε ζητήσει το λόγο. Ναι, μια ερώτηση έχω να κάνω κι εγώ. Μα είπατε ότι πρέπει να μειωθεί το κόστο τη ε, τυποποίηση. Βέβαια, αυτό αφορά το συνολικό κόστο τη παγκοσμιοποίηση. Πώς αξιολογείται το κόστος και τις δυσκολίες σε σχέση με συγκεκριμένες χώρες. κόστος μείων φόρος που πληρώνει η αμυντική βιομηχανία. Μπορείτε να μας πείτε πώς το αξιολογείτε αυτό αναχώρα. για την επέκταση τώρα. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 28 κρατών μελών. Το κάθε κράτο μέλο μπορεί να έχει να μην έχει κάποια υποδομή. Εξαρτάται και από τις πολιτικές μας. Η πολιτική μας ε, επηρεάζει τα δημοσιονομικά μέσα που έχουμε. Αλλά αυτή, αυτά τα μέσα δεν είναι πάντοτε στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο. Αυτά τα καλά αποτελέσματα πώς μπορούμε να τα καταστήσουμε έτσι κάπως ε, πιο οικουμενικά. Thank each one of them um, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για το θέμα της απαξίωσης των παροχημένων και κατά πόσο μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι εδώ. Ένα σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν κοιτάμε την αμυντική βιομηχανία στις πρώτες φάσεις είναι ότι οι θεσμοί δεν παίζουν και τόσο σημαντικό ρόλο σε σχέση με τα πρότυπα που θα πρέπει να αναπτυχθούν για το μέλλον. Γιατί μιλάμε για συστατικά και στοιχεία στα οποία αυτές οι μηχανίες είναι πρωτοπόρες. Και είναι από αυτούς που ζητούν την θέσπιση Γι' αυτό ακριβώς τόνισα την σημασία των βάσεων των δεδομένων που έχουμε. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση της χρήσης και από τι και από τη βιομηχανία, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για πρότυπα για την πολιτική και αμυντική βιομηχανία, τότε θα πρέπει να καθοδηγεί, να ηγείται η βιομηχανία ίδια. Γιατί είδαμε στις μελέτες ότι οι ενόπλες δυνάμεις, οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι θεσμοί παρόλο που έχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μείωση του κόστους και την αύξηση της διαλειτουργικότητας παραδοσιακά. Πώς να το πω αυτό. Δεν είναι και τόσο καλή στο να κατανοήσουν την προέλευση των τεχνολογικών εξελίξεων και που βρίσκονται τα όρια, τα σύνορα της τεχνολογίας. Γιατί συνήθως αυτό, σε αυτό είναι καλύτερη η βιομηχανία και η αμυντική βιομηχανία, μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Και όπως είπατε και εσεί σωστά, και εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν τεράστιο ρόλο στην καινοτομία. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και ξανατονίζω, να εμπλακεί πολύ περισσότερο μηχανία από ό,τι μέχρι τώρα. Τώρα για τη στρατιωτική κινητικότητα. Παρά το γεγονό ότι ένα από τα κύρια συνεργασία συνεργασίας Ένωση θα έλεγα την πλευρά της Ένωσης, παρόλο που είχαμε μία πρόταση για 6,5 δις στο ΠΔΠ, στο πρόγραμμα αυτό, υπάρχει μια ευκαιρία για την Ένωση, επειδή οι επενδύσεις, το μεγαλύτερο τμήμα της επένδυσης αυτής θα είναι διπλής χρήσης, δηλαδή υπάρχουσες υποδομές και μεταφορές ε, δυναμικού και υποδομών στρατιωτικών η διαφορά είναι ότι καμιά φορά αυτή η απόκληση μεταξύ της ανάγκης για υποδομές και της συμφωνίας για τις στρατιωτικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δική μας διαδικασία εντοπισμού των αναγκών. Η δυσκολία προκύπτει από το να τα μεταφέρουμε όλα αυτά στο ΝΑΤΟ. Η πρόταση διακόπτη, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι άμεσα θα σταματήσει η διερμηνία και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά χωρίς διερμηνία. Ε, στο συγγνώμη ήταν δύσκολη ημέρα σήμερα, είναι αλήθεια, με πολύ μακροσκελείς εισηγήσει. Ωραία, τότε να είμαι πολύ σύντομο σε περίπτωση που έχουμε και ερωτήσεις. Έχουμε λοιπόν για τη στρατική κινητικότητα την ανάγκη να τονίσουμε ότι οι τρονές υποδομές αφορούν βεβαίως τους ε, πολιτικούς στόχους, αλλά ε, υπάρχει ένα κομμάτι στρατιωτική κινητικότητα. Έχουμε λοιπόν αυτέ τι ανάγκε οι οποίε απορρέουν από το ΝΑΤΟ, από ΝΑΤΟ και, έχουμε και τι ίδιε τι ανάγκε τη Ένωση όσον αφορά τη στρατιωτική χρήση. Βεβαίω, οι χώρε μέλη βεβαίω ε, είναι αυτέ που αναπτύσσουν τι υποδομέ αυτέ. Τώρα, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γι' αυτό ακριβώ το λόγο έχουμε φτιάξει αυτό το εργαλείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα η διαφορά είναι βέβαια ότι στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνα βλέπουμε ότι η βιομηχανία επικεντρώνεται κυρίω ή συγκεντρώνεται κυρίως κυρίω σε κάποιε χώρε μέλη. Έχουν μεγάλε επιχειρήσει οι οποίε ε, ε, παρέχουν ή τροφοδοτούν τις διάφορες χώρες. Τώρα το δίλημα είναι ότι έχουμε ένα κατακαιρματισμό στις εθνικές γραμμές εφοδιασμού, αλλά το θέμα είναι πώ θα μπορούσε κανεί σε αυτό το πλαίσιο να μην παραβλέψει την καινοτομία. Και εκεί ακριβώς θα πρέπει να δούμε πώς η καινοτομία θα μπορούσε να προσέλθει και από τις μικρομεσαίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα βέβαια, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω πολύ σύντομα κάποια από αυτά. Καταρχάς, το κεφάλαιο που είναι διαθέσιμο για την έρευνα και τη τεχνολογία. κεφάλαιο που είναι συνήθως χαμηλά, επειδή προσπαθούν να αναπτύξουν πρωτότυπα σε επαγγελματικό επίπεδο